Σα Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της διάταξη και περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι η κοινή συνεδρία με το της δημόσιας υγείας και ασφάλισης των τροφίμων. ορίσω τους συναδέλφους, ε, την Ένβη. Συγγνώμη που καθυστερήσαμε λίγο. Ήρθε και η πρόεδρος, κύριε Βαλεάν. Καλώς ήρθατε. Πρώτο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων παρουσία της Κομισιόν ε, για την παρακολούθηση και εντοπισμό των προϊόντων καπνού. Περιμένουμε και μια κατεξοδότηση πράξη στο τέλος του χρόνου για αυτό το θέμα ε, σε ό,τι αφορά την είσοδο αδασμολόγητων προϊόντων, πώς μπορούμε να εντοπίζουμε την είσοδο τέτοιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, περιμένουμε και με βάση τα άρθρα 15 και 16 την ε, εφαρμογή ε, του σχετικού κανονισμού για τα προϊόντα καπνού μέχρι το τέλος του χρόνου με τις κατεξοδοτήσεις πράς, πάρα πολύ σημαντικές κατεξοδοτήσεις πράξεις. Γι' αυτό οργανώσαμε και αυτή τη συνάντηση σήμερα γιατί θέλουμε να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης ε, και εντοπισμού των ε, προϊόντων. Έχουμε και τις ε, διατάξεις του πρωτοκόλου της ΠΟΗ που πρέπει να στηρίξουμε, να εφαρμόσουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν σε αυτούς του, να υπάρχει αυτό το unique identifiers Πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Το 80% των παράνομων προϊόντων έρχονται εκτός από αγορές εκτός Ένωσης και τα πιο πολλά είναι τα λεγόμενα παράνομα λευκά, τα πακέτα χωρίς διακριτικά δηλαδή και τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να κατάσχουμε. Ε, αναμένεται ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι και στο εμπόριο και στη βιομηχανία και οι μικροί λιανοπολιτές και οι χονδικοί φοβούνται τι θα γίνει με αυτό το νέο σύστημα. Μήπως επηρεάσει και τις εμπορικές δομές, ε, ιδίως ε, στην Ήπεθρο. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα που θα είναι αποδοτικός προς το κόστος, θα είναι ένα ανοιχτό σύστημα, να αποφύγουμε δηλαδή τα μονοπόλια γιατί όλα αυτά συνδέονται με τεράστιο κόστος. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα παγκόσμιο πρότυπο, ένα παγκόσμιο κανόνα. Και φυσικά όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα ήρθαν με το ένα τεράστιο λόμπι, γιατί πραγματικά είναι όλα αυτά που διακυβεύονται. Θέλουμε να έχουμε λοιπόν ένα ανοιχτό σύστημα, ε, που όμως δεν μπορεί να περιλάβει τα στοιχεία των προηγούμενων συστημάτων. Έχουμε προσκαλέσει δύο ε, εμπειρογνώμονες. Έχουμε και εκτός από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΕ και όλα την κυρία Μπερτελέτη και Διευθύντρια της Mock Free Partnership και τον κύριο ε, Λεκέν. Η κυρία Μπερτελέτη που είναι όμως, γιατί δεν τη βλέπω. Α, είστε έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Σας ε, καλωσορίζω και τον Λεκέν φυσικά θέλω να καλωσορίσω. Ερικ Λεκέν, Center of Competence Track and Trace. Ένα ε, κέντρο που προτείνει λύσεις, έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα ιχνηλασιμότητας εντοπισμού ε, προϊόντων καπνού και σε άλλους ρυθμισμένους τομείς όπως είναι τα φάρμακα, τα τρόφιμα, τα εξαρτήματα μηχανημάτων. Θα δούμε λοιπόν και τι έχει να μας πει για το track and trace των προϊόντων καπνού. Πώς λοιπόν έχουν εξελιχθεί μέχρι τώρα τα πράγματα, ποιες είναι οι προσδοκίες, καλύπτονται αυτά που θα έχουμε ζητήσει. κυρία Βαλεάν, μπορείτε να ξεκινήσετε στην την τη της συζήτησης. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να σας καλυξορίσω σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού για τον και τον Εντοπισμό των Προϊόντων Καπνού. Οι δύο επιτροπέ αποφασίσαμε να καλέσουμε σημαντικού ομιλητέ για την ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το πάνελ θα μας δώσει την ευκαιρία, πιστεύουμε, να συζητήσουμε ένα θέμα ζωτικής σημασίας ε, για να διαφυλάξουμε την υγεία των Ευρωπαίων. Αυτό είναι ο σκοπός μας και αυτό θέλουμε να προκύψει από αυτή τη συζήτηση, γιατί αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε. Φυσικά θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα για το πώς αυτό το νέο πλαίσιο θα βοηθούσε την καταπολέμηση ε, των παράνομης ε, παρασκευής ε, και το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού. Γιατί πρόκειται για κίνδυνο δημόσιας υγείας, όπως υπόθηκε και από την πρόεδρο Γκρέσλε. Έχουμε σημαντικούς όγκους παράνομων προϊόντων που δεν πληρούν τις ε, προϋποθέσεις ε, της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού, κυκλοφορούν στην αγορά και υπάρχει ένδειξη ότι μπορεί να αυξηθούν οι όγκοι αυτοί. Επομένως, ανησυχούμε ότι αυτά τα παράνομα προϊόντα θα υποσκάψουν ε, την κυκλοφορία των νόμων προϊόντων και την προστασία που προβλέπεται από την νομοθεσία. Αυτό είναι λυπηρό και είναι σημαντικό να έχουμε ένα επιτυχές και πλήρες πλαίσιο που να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Φυσικά, πρέπει και εμείς να κατανοήσουμε πώς ακριβώς μπορούμε να συνεισφέρουμε στην καταπολέμηση των παράνομων προϊόντων στην αγορά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τα ακούσουμε όλα αυτά. Λεφτέντων αυτών, εν συντομία. Γιατί έχουμε ήδη τους ανθρώπους εδώ που γνωρίζουν τα θέματα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σέσελ ε, ο οποίο ε, είναι αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, εξαιτήμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, σα ευχαριστώ που με καλέσατε να μιλήσω εκ μέρου τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΑ για την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα τη χρησιμότητα και εντοπισμού των προϊόντων καπνού. Η Κομισιόν εργάζεται για την εφαρμογή ενός νέου συστήματος χρησιμότητας και του για τα προϊόντα καπνού, όπως προβλέπετε από το άρθρο 15 της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. Χαίρομαι λοιπόν που έχω την ευκαιρία να σας δώσω μια επικαιροποίηση για το έργο αυτό και επίσης να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Κομισιόν. Καταρχήν όμω, θα ήθελα να επενθυμίσω τον κύριο στόχο που δημιουργήσαμε ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και του λόγου που συμπεριλαμβάνουμε τέτοιε διατάξει στην οδηγία το παράνομο εμπόριο καπνού έχει ε, σοβαρό επιζήμιο αποτέλεσμα στην κοινωνία. Καταρχήν ε, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών καθώς δίνει πρόσβαση σε πιο φτηνά προϊόντα καπνού τα οποία ε, δημιουργούν και διατηρούν τον εθισμό κυρίως σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως είναι η δεύτερον υποσκάπτει τις καλύτερες προσπαθίες μας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Τα παράνομα προϊόντα καπνού είναι πολύ λιγότερο πιθανό να σέβονται τις βασικές απαιτήσει ε, του κανονισμού ως προς τα συστατικά και τις προειδοποίησεις ε, για την υγεία. Βαρλεμάντος στην οδηγία. Αυτός ο κανονισμός ε, ε, ουσιαστικά ε, προσπαθεί να αποτρέψει τους νέους ανθρώπους από την κατανάλωση καπνού και πρέπει να αναφέρω και τα τεράστια ποσά που χάνονται ετησίως από τις κυβερνήσεις ως αποτέλεσμα της παράνομης αυτής δραστηριότητας. Και εκτιμάται ότι είναι περίπου 11 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό φυσικά πλήττει τους εθνικούς προπολογισμού και τροφοδοτεί το οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει λοιπόν λόγο να δράσουμε και νομίζω ότι ακούσαμε ξεκάθαρα αυτό το μήνυμα στην Κομισιόν από την αρχή και γι' αυτό το λόγο θέσαμε ως προτεραιότητα την εφαρμογή του πρωτοκόλου FCTC της Σύμβασης Πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού για να εξαλειψούμε τα παράνομα προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι ε, σέβεται το πρωτόκολλο όταν το, το τον Ιούνιο του 2016 και θέλουμε να προωθήσουμε την επικύρωσή του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς προκειμένου να τεθεί γρηγορότερα σε ισχύ το πρωτόκολλο. Η κύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε σαφές μήνυμα στους διεθνεί εταίρους ότι ε, ε, θέλει να καταπολεμήσει το παράνομο εμπόριο και ε, ουσιαστικά προετοιμάζει το δρόμο για τη συγκεκριμένη εφαρμογή του. Και ε, εδώ έρχεται και το σύστημα χρηματισμότητας και εντοπισμού. Το άρθρο 15 της ε, οδηγίας για τα προϊόντα καπνού θα δημιουργήσει ένα εξάρτητο σύστημα χρηματισμότητας για όλα τα προϊόντα καπνού που παράγονται ε, και προορίζονται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου FCTC θα εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΓΑΜΑ είναι αρμόδια εντός της Κομισιόν σε στενή συνεργασία με τους συναδέλφους στην ΟΛΑΦ και στις άλλες υπηρεσίες και είναι υπεύθυνη για να δώσει δευτερογενή νομοθεσία που είναι απαραίτητη για να λειτουργήσει πλήρω το σύστημα. Σα διασφαλίζω ότι είναι υψηλή προτεραιότητα για την Κομισιόν αυτό το project και εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτό το καθήκον. Είναι βέβαια και πολύπλοκο καθήκον να έχει τεχνικό, στρατηγικό και μακροπρόθεσμο προβληματισμό, ένα και φιλόδοξο με εξαφή νομική προθεσμία για την εφαρμογή του συστήματο, το οποίο υπάρχει στην οδηγία 20 Μαου 2019. Όμως ε, είμαστε εντός του χρόνου και είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να σεβαστούμε τον ενδυτικό σχεδιασμό μας. Η κύρια προτεραιότητά μα είναι ένα σύστημα που να λειτουργεί, να είναι αποτελεσματικό, να καταπολεμεί το παράνομο εμπόριο στο προϊόντα καπνού και να διασφαλίσει την αλυσίδα ε, προμήθειας, αλλά και να προστατεύσει τη δημόσια υγεία βάσει του υφισταμένου κανονισμού. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα που να αντιμετωπίζει τις πραγματικότητες, την πραγματικότητα της και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει μια διαβούλευση ε, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουμε δημόσια διαβούλευση, έρευνες στην αγορά, καθώς και συναντήσεις ε, προσωπικές με, τους, ε, με τα ενδιαφερόμενα μέρη για να έχουμε τεχνική και πολιτική συνεισφορά από τα ενδιαφερόμενα μέρη και της ΜΚΟ σε ό,τι αφορά τη δουλειά της εφαρμογής. Σε όλα αυτά η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΤΕ έχει σεβαστεί πλήρως τις υποχρεώσεις της Σύμβασης Πλαισίου ε, και έρχομαστε σε επαφή με την καπνοβιομηχανία μόνο την απαραίτητο για να ε, δημοσιεύσουμε και, δημοσιεύουμε και τα πρακτικά των συζητήσεων. Επίσης, ε, τακτικά συναντούμαστε για να διασφαλίσουμε ότι οι ανάγκες των Διεκτικών αρχών θα καλύπτονται από το σύστημα. Ε, θα ε, πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα εχνηλεσιμότητας και εντοπισμού και τα μέτρα του φυσικά πρέπει να είναι ανάλογα του στόχου και θα πρέπει να έχουν κατά νου και τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα μέτρα που θα προτεθούν σίγουρα θα το πετύχουν αυτό και θα μα δείξουν ότι είναι και αποτελεσματικά ω προ το κόστο. Ένα άλλο ξεκάθαρο κριτήριο για την αποτελεσματικότητα θα είναι η πλήρη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο τη Σύμβαση Πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού και ε, τι απέτηση να διασφαλίσουμε ότι το σύστημα εχνηλασιμότητα είναι σε πλήρη έλεγχο από τι αρχέ. Αυτό είναι υψηλή προτεραιότητα από την αρχή για την Κομισιόν και όλε οι πολιτικέ, όλε οι επιλογέ πολιτική ελέγχονται για να το πετύχουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, έχουμε ένα ενεργητικό σχεδιασμό που προβλέπει την υιοθέτηση των σχετικών πράξεων μέχρι τα τέλη του έτου. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑΣΑΝΤΗ επίση κατάρτισε ένα εσωτερικό σχεδιασμό λεπτομερή και όπω σα είπα θα το σεβαστούμε. Συνεχίζουμε την πρόοδο με τι εσωτερικέ μα διαδικασίε καθώ και με τι συζητήσει με τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε ότι το σχέδιο τη νομοθεσία θα δημοσιευτεί για διαβούλευση το καλοκαίρι σύμφωνα με το θεματολόγιο καλύτερη νομοθεσία. Πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν διακυβεύεται εδώ μόνο το ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά μπορεί και άλλα μέρη θα στραφούν στο μοντέλο χρησιμότητας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα εφαρμόσουν τα συστήματα του στο μέλλον, καθώ και τι λύσει που θα επιλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είναι πιο επιτακτικό να διασφαλίσουμε ότι τα υψηλά πρότυπα συμμόρφωση και αποτελεσματικότητα στήθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτές ε, οι σκέψεις ε, υπήρχαν ε, στο πνεύμα της ε, Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας ε, σήμερα. Το Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ευαισθητοποίηση, για τη σημασία να υπάρχει καλή εφαρμογή του πρωτοκόλλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευχαρίστω στα απαντήσω σε ερωτήσεις που έχετε σε σχέση με τα όσα σας εξέθεσα εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάργκρετ Χόφμαν, Διευθύντρια παρακαλώ.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 Ευχαριστώ πολύ κυρίες Πρόεδροι, σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στη συνάντηση αυτή που είναι πολύ σημαντική. Για μία ακόμα φορά θέλω να ξεκαθαρίσω. Θα γνωρίζετε ότι είναι μια, η Όλαφ είναι Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η ρυθμόν ένα επιτροπή που ε, ε, αντιμετωπίζει τις ε, παράνομες πωλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επίσης ε, οι συνάδελφοι ασχολούνται με την υλοποίηση του συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού. Έτσι βρισκόμαστε όλοι εδώ ως υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πετύχουμε την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Αναγνωρίζουμε ως όλα την σημασία αλλά και τις δυσκολίες του έργου των συναδέλφων της Επιτροπής για να εξισορροπηθούν οι ανάγκες πολλών εμπλεκομένων και τις απαιτήσεις και να καταλήξουν σε ένα, καλά, ε, σε ένα εύρυθμο σύστημα παρακολούθησης και λειτουργίας. Ε, αυτό έχει ήδη συζητηθεί. Αυτό που θα ήθελα σήμερα να κάνω εδώ, γιατί όπως σας είπα στην αρχή είμαστε η επικεφαλής υπηρεσία για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, προϊόντων καπνού, ήθελα να ε, θέσω ε, τη συζήτηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να σας πω πού βρισκόμαστε όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζουμε για την καταπολέμηση του παράνομης εμπορίας καπνού. Ξέρετε ότι είναι μια διαρκής δυσκολία και το επίπεδο παράνομων πωλήσεων είναι απαράδεκτα υψηλό είναι απαράδεκτο αυτό και από άποψη υγείας, από άποψη δημοσιονομική και από άποψη ασφάλειας. Θα γνωρίζετε ότι το 2013 η Κομισιόν ε, υιοθέτησε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ε, αύξηση της ε, ε, ενίσχυσης καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου. Είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα το 2013. Ήταν αρκετά ενθαρρυντικές οι προτάσεις σε ένα πρόγραμμα δράσης με 50 δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών μελών. Τώρα ε, ε, ουσιαστικά έχουμε ολοκληρώσει την υλοποίηση του προγράμματος δράσης. Ενδεχομένως θα γνωρίζετε ότι έχει σταλεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Ε, Κάναμε μελέτη για την προόδο αυτής της στρατηγικής του 2013 και φέτος ε, το Μάιο ε, υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λεγόμενο Tobacco Implementation Report που απευθύνεται στα θεσμικά όργανα και ανακεφαλαιώσαμε ε, τα βασικά ζητήματα της έκθεσης αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, έναν απολογισμό της πρόοδου από το 2013 και επιπλέον, αυτό που είναι πιο σημαντικό υποθέτω και για σας, παρουσιάζουμε κάποιες ιδέες για μελλοντικές δράσεις. Τα ευρήματα της έκθεσής μας είναι εν σε επίπεδο κρατών μελών και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως Όλαφ ε, επιτύχαμε το στόχο μας για την ε, ενίσχυση της καταπολέμησης των παράνομων ε, πολίσεων και από άποψη δίωξης. Παραδείγματος χάρη οι κατασχέσεις παράνομων τσιγάρων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά ένα πέμπτο από το 2013 από 3,1 δις σε 3,8 ε, δις τσιγάρα. Όλα αυτά η Όλαφ συμμετείχε και στις έρευνες αλλά και στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης όσον αφορά τα έσοδα. Έχουμε 1,1 ε, δις εκατομμύρια τσιγάρα που κατασχέθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. Τώρα, στον τομέα της πολιτικής, όπως είπε και ο Μάρτιν, τα βασικά στοιχεία της εφαρμογής της στρατηγικής και του προγράμματος δράσης ήταν η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά και με την οδηγία για τα προϊόντα καπνού και με την υπογραφή και κύρωση του πρωτοκόλου FCTC. Και ε, είμαστε ευγνώμονες στο Κοινοβούλιο που το υποστήριξε και έγινε και ε, το κύρωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2016 και πάλι ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή σας. Παρά τα αυτά, πρέπει να παραδεχτούμε ότι αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο, κυρίως όσον αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό, δεν έχει τεθεί ισχύ. Το πρωτόκολλο FCTC δεν εφαρμόζεται. Έχουμε 16 κυρώσεις, χρειάζονται 40 και που πρέπει να πρέπει να γίνουν 40, μόνο 6 κράτη-μέλη έχουν, το έχουν κυρώσει. Όπως είπε ο κύριος Μισελ, πρέπει, πρέπει να προωθηθεί ενεργητικά στα κράτη-μέλη αυτή η κύρωση. Επίσης και σε σχετικές τρίτες χώρες να γίνει αυτή η προώθηση. Νομίζω ότι δίνεται μια όθηση στις συζητήσεις και ελπίζουμε ότι θα έχει κυρωθεί πριν από το 2018. Παρά τα αυτά πρέπει να υπογραμμίσω ότι για να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό το πρωτόκολλο με αποτελεσματικές διατάξεις χρειαζόμαστε να συμμετέχουν οι βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης. Αυτό είναι σημαντικό για τις διατάξεις παρακολούθησης και εντοπισμού. Και όπως ήδη ακούσαμε, ε, όταν υλοποιηθούν οι διατάξεις ε, της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού θα εφαρμοστούν και οι σχετικές διατάξεις του πρωτοκόλου FCTC. Συνολικά λοιπόν έχει γίνει προόδος στον τομέα της ε, δίωξης και το νομοθετικό τομέα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες, όπως όμως όλοι γνωρίζουμε, η παράνομη αγορά ε, συνεχώς ε, αλλάζει, όπως είπατε και εσείς έχουμε το φαινόμενο των cheap whites, των φθηνών λευκών τσιγάρων, ε, που έχει αναφερθεί και στη στρατηγική του 2013. Έχουμε λοιπόν τα νέα, ε, να προσαρμόζουμε, την ανάγκη να προσαρμόζουμε τα εργαλεία μας στις νέες προκλήσεις. Έχουμε το ψήφισμά σας του Μαρτίου 2016 και η Επιτροπή ε, εσωτερικά αντιμετωπίζει το θέμα μετά την ε, έκθεση του Tobacco Implementation Report του Μαΐου για να προσπαθεί να ενισχύσει τα μέσα της και να προσθέσει νέα. Δεν μπορώ επ' αυτού να προσθέσω ε, τίποτα ακόμα γιατί εξακολουθούμε να το... Ε, μελετάμε το θέμα. Ακούσαμε όμως από την Εστονική Προεδρία ότι θα υποβάλουν συμπεράσματα του Συμβουλίου για την έκθεση αυτή του Μαΐου και επίσης είναι ευπρόσδεκτη η ε, προσφορά, η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με βάση τις διαβουλεύσεις αυτές του με το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και τους άλλους εμπλεκόμενους περιμένουμε ότι η Κομισιόν θα παρακολουθήσει την συνέχεια της, έκθεση, της έκθεσης εφαρμογής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Παρτελέτη έχει τώρα το λόγο. Μπερτελέτη. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Of... Ευχαριστώ. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Κατά την παρουσίαση αυτή θα σας ε, εξηγήσω τι είναι η εταιρική σχέση Smoke Free Partnership και πώς λειτουργούμε. Και θα ήθελα να δηλώσω επίσημα ότι ποτέ δεν έχω λάβει καμία χρηματοδότηση από εμπορικές οντότητες που έχουν συμφέρον ε, για τις συζητήσεις, ε, για τα αποτελέσματα της, ε, των ευρωπαϊκών συζητήσεων ή της FCTC. Επίσης, θέλω να τονίσω επίσημα ότι δεν είμαι εμπειρογνώμονας στην τη της και στον εντοπισμό, όμως κατανοώ το, στόχο του, το σκοπό του. Έτσι λοιπόν, ε, ε, συντομία, ο συνασπισμό ε, Smoke Free Partnership είναι ένα μεγάλο δίκτυο που τελείται από 42 οργανώσεις σε 22 χώρες και έχουμε εταιρικέ σχέσεις με τρεις διεθνείς οργανισμούς παγκόσμιας εμβέλειας. Κάνουμε αυτά που κάνουμε γιατί όπως ακούσαμε η κατανάλωση του καπνού παραμένει η μόνη μεγαλύτερη αιτία θανάτου που μπορεί να αποφευχθεί στην Ευρώπη και αυτός ε, είναι ο κύριος κίνδυνος για καρδιακές ε, ασθένειες, αναπνευστικές ασθένειες και τα λοιπά που μπορεί να, να αποφευχθεί. παράνομη πώληση προϊόντων καπνού ε, χρησιμοποιείται για να υποσκαφτούν τα μέτρα ελέγχου του καπνού, να διαδοθεί η επιδημία του καπνίσματος και να υπάρχουν και πώληση εισόδων για τις κυβερνήσεις. Τι σημαίνει κάποιος ε, να βλέπει το δέντρο και όχι το δάσος από την αρχή των διαπραγματεύσεων όλοι επικεντρώθηκαν υπερβολικά ε, στις λεπτομέρειες του συστήματος συχνηλασιμότητας και τοπισμού. Είχαμε μία συνάντηση ενδιαφερομένων μερών. Το σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο και αν και ακόμα όλα έχουν γίνει είναι αυτές προσπάθειες ε, να εξηγηθεί πώς θα μοιάζει το σύστημα ειχνηλασιμότητας και τοπισμού, φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι πολίτες ε, θα χαθούν στη μετάφραση. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα εδώ, βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Διάλεξα αυτή την έκφραση γιατί σημαίνει ότι αν επικεντρωθεί πάρα πολύ στις λεπτομέρειες και στην πολυπλοκότητα ενό στοιχείου μπορεί να χάσεις τη μεγαλύτερη εικόνα ή το σημαντικό σημείο. Όπως σα είπα, δεν είμαι εμπειρογνώμονα στην χρησιμοποιώ και εντοπισμό, Ούτω ή άλλως, επομένως ε, θα επικεντρωθώ στο δάσο, στην παρουσίασή μου. Ε, θα ήθελα ίσω ε, να Ρίξτε και εσείς μια ματιά μαζί μου και να ανακαλύψουμε το δάσος. Θέλουμε να δούμε τη συνολική εικόνα και τις κύριες πτυχές αυτού του φακέλου. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που θα πρέπει να θέσουμε στον αυτό μας είναι η εξής. Ποιος είναι ο σκοπός ενός συστήματος συμφιλεσιμότητας και εντοπισμού. Εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο σύστημα για προϊόντα καπνού θα πρέπει να επιτρέψει στις ελληνικές αρχές να ελέγχουν και παρακολουθούν τα προϊόντα καπνού στην αλυσίδα εφοδιασμού. Επίσης το σύστημα πρέπει να ε, διευκολύνει τον εντοπισμό του σημείου στην αλυσίδα όπου προϊόντα καπνού που έχουν παρασκευαστεί νόμιμα διοχετεύονται στην παράνομη αγορά. Και θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα εδώ πρέπει να πούμε ότι καταβλήθηκαν οι δασμοί, παραδείγματο χάρη το 2014, η, ε, επιβλήθηκε ε, ένα πρόστιμο στην British American Tobacco από το Βέλγιο, γιατί είχε διοχετεύσει παράνομα προϊόντα στην αγορά. Αυτό σημαίνει ότι η καπνοβιομηχανία εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την λαθρεμπόριο το δικό της προϊόντων. Ίσως θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν. Επομένως, θα πρέπει να δούμε τι συνέβη στο παρελθόν και να ξεκινήσουμε από πού ξεκινήσαμε. Τον Νοέμβριο του 1999 η Καναδική κυβέρνηση μήνυσε την καπνοβιομηχανία στα Αμερικανικά δικαστήρια όταν προέκτησαν αποδεκτικά στοιχεία για λαθρεμπόριο από την καπνοβιομηχανία. Το Μάιο του 2000 ε, κάποιοι κολομβιανοί κυβερνήτε επίση μήνυσαν τη Φίλιπ Μόρι στα Αμερικανικά δικαστήρια για λαθρεμπόριο τσιγάρων και τον Νοέμβριο του 2000 η Ευρωπαϊκή Ένωση και 10 κράτη-μέλη άσκησαν μήνυση κατά της Φίλιπ Μόλι, της Japan Tobacco International και της J.R. Reynolds και την κατηγόρησαν ότι σκόπευαν ε, να προβούν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων και να θα ρυθμίσουν τις τιμές, να δωροδοκίσουν δημόσιους αξιωματούχους και ε, ουσιαστικά να κάνουν παράνομο εμπόριο, ε, χρηματοδοτώντας και τρομοκρατικές ομάδες. Τώρα, αυτό Ευ- την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει επικεφαλής των διαπραγματεύσεων προς ένα διεθνές ε, πρωτόκολλο κατά του λαθρεμπόριου καπνού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, ουσιαστικά επικεφαλής αυτών των διαπραγματεύσεων και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι. Επομένως, μπορεί να πει κανεί ότι αυτό ήταν ε, στο παρελθόν. Τι συμβαίνει στο παρόν. Έριξα μια ματιά σε ένα σημείωμα τη 28η Ιουνίου, πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα, που γράφτηκε από την Προεδρία, στέλνει από την Προεδρία στην υψηλή ομάδα εργασία, στην ομάδα υψηλού επίπεδου των Γενικών Διευθυντών για τα Τελωμία και λέγεται ότι το ελευθερεμπόριο από του ε, μεγαλύτερου παραγωγού σήμερα ε, δεν λαμβάνει τόσο μεγάλο μέρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη πλευρά, τα φτηνά λευκά πακέτα ε, και τα λαθρέα τσιγάρα σήμερα κυριαρχούν ε, στις μεγάλες κατασχέσεις. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε στοιχεία από το 2011 και το 2012 είναι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνίων και μας δείχνει ότι το ελευθερμπόριο γνήσιων τσιγάρων είναι αρκετά υψηλό. Πολύ υψηλότερο από ό,τι τα φτηνά λευκά πακέτα και τα παραπημένα τσιγάρα. Εδώ είναι κάπως ε, αστείο αυτό το, κάπως περίεργο αυτό το slide, αυτή η διαφάνεια προέρχεται από μία παρουσίαση της PMI στους μετόχους της ε, και λέγεται ε, ότι το 2013 από όλα τα τσιγάρα που πουλήθηκαν στην Κίνα μόνο το 2% ε, ήταν ε, λαφρέα τσιγάρα. Ίσως να έχει διαφορετική αφήγηση η καπνοβιομηχανία. Είδαμε όμως ε, στο προηγούμενη διαφάνεια ότι έχουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, μπορεί να πείτε ναι, αυτά είναι αριθμητικά στοιχεία, αλλά τα αριθμητικά στοιχεία από τον κόσμο, από τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για να δούμε στη συνέχεια. Εδώ έχουμε μία σύνοψη των διάφορων εκθέσεων της Project Sun και εγώ από ό,τι κατάλαβα βλέπετε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δείχνει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούμε να έχουμε 56% της παράνομης αγοράς που σχετίζεται με γνήσια τσιγάρα σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της καπνοβιομηχανίας. Έτσι λοιπόν, όποια δεδομένα και δούμε, είτε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια, μπορούμε να δούμε παρόμοια αποτελέσματα, ότι πάνω από το ίμιση της παράνομης αγοράς είναι προϊόντα που προέρχονται από τις καπνοβιομηχανίες. Έτσι λοιπόν, ε, ίσως ε, οι καπνοβιομηχανίες ε, ε έκαναν ε, μια ιστορία καταστροφής, ε, μια ιστορία επιτυχίας, όπου παρουσιάζονται να είναι και θύματα, αλλά και μέρος της λύσης. Όμως έχουν αλλάξει τα αποδεικτικά στοιχεία και έχει αλλάξει και η φύση των παράνομων προϊόντων και σήμερα δεν μας πείθει τόσο η ιστορία της καπνοβιομηχανίας. Ποια ήταν ε, η στρατηγική της καπνοβιομηχανίας, Θέλω να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είναι καθαρή στο παρελθόν, τα τελευταία δέκα χρόνια, η καπνοβιομηχανία παρουσίασε τις προσπαθίε τη ω παραδείγματα συνεργασία και διασφάλισε ότι οι διοκτικές αρχές θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα παραχάραξης και ανταγωνισμού από μικρούς παίκτε, δηλαδή από τα φτηνά λευκά και ανέπτυξαν το δικό τους σύστημα, το Contentify, ως μια πλήρη λύση για το παράνομο εμπόριο. Το Contentify έχει το πλεονέκτημα να κρατά Τη κυβερνήσεις έξω από τα εργοστάσια και να θέτει την καπνοβιομηχανία ω κύριο εταίρο στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Τουλάχιστον έτσι όπω περιγράφηκε τουλάχιστον δημοσίω το σύστημα Contentify δεν μας δίνει κανένα τρόπο να ξέρουμε ποιο κωδικό είναι γνήσιο, ακόμη και αν ε, ανακαλύψουμε ε, ουσιαστικά παράνομα προϊόντα. Έτσι λοιπόν ε, κάλυψε τα ίχνη της ε, η καπνοβιομηχανία, πούλησε τον Contemptify σε ανεξάρτητες εταιρείε. και πραγματικά τα πάνε πάρα πολύ καλά πουλώντας τον Contemptify σε φερόμενες ανεξάρτητες εταιρείε. Έτσι λοιπόν σήμερα ποιος προωθεί τη λύση της καπνοβιομηχανίας, μπορείτε να μας πείτε ποιος μπορεί να το πει αυτό. Παραδείγματο χάρη, ενώ ο κύριος Λεκένο εδώ δίπλα μου παρόν μπορεί να φαίνεται ανεξάρτητος σε εσάς, έχει προωθήσει ποτέ το Contentify στο παρελθόν, έχει κάνει παρουσιάσεις, άρθρα, έχει συμμετέχει σε διάφορες συναντήσεις για να υποστηρίξει το Contentify και αν το έκανε θα εμπιστευόταν τη λύση που θέλει να προωθήσει. Είναι απλώς ερωτήσεις αυτές. Θέλω να κλείσω, γιατί νομίζω ότι φτάνω και στο πλήρωμα του χρόνου. Θα ήθελα να πω ότι η καπνοβιομηχανία εξακολουθεί να εμπλέκεται στην παράνομη εμπορία προϊόντων και ακόμη και είναι αλήθεια ότι έχουμε λιγότερες κατασχέσεις. Αν έχετε μια περικαλιά στο σπίτι σας και βάλετε ε, το συναγερμό και δεν υπάρχει φωτιά, τι θα κάνετε, θα αφαιρέσετε το συναγερμό επειδή τέλος πάντων δεν ξέσπασε πραγματική πυρκαγιά, το σύστημα υπάρχει για να ελέγχει την αλυσίδα εφοδιασμού των δικών τους προϊόντων και ακριβώς ε, αυτό θα έπρεπε να είναι και ο σκοπός του συστήματος Tracking and Trace. Το παράνομο εμπόριο, όπως ακούσαμε, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και χρειάζεται παγκόσμια λύση. Και ε, πράγματι το πρωτόκολλο της Σύμβασης Πλησίου για τον Ελέγχο του Καπνού είναι η απάντηση, οποιαδήποτε οργάνωση που προωθεί το σύστημα Contentify ε, ουσιαστικά θα πρέπει να διενευνηθεί και θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσουν ότι ένα τρίτο μέρο εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το σύστημα, ελέγχει το σύστημα για να είναι σίγουρο ότι οποιαδήποτε κατάχρηση από την καπιοβιομηχανία ε, έχει αφαιρεθεί. είχα δώσει κάποιες ιδέες ε, σε σχέση με τα δέντρα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο ορισμός της ανεξαρτησίας είναι στεγανός ε, και απελευθερωμένος από καπνό στο σύστημα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι συμβάσεις μεταξύ των ε, καπνοβιομηχάνων και των εταιριών αποθήκευσης των δεδομένων μπορεί να ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την υπογραφή της σύμβασης. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και το νέο αναγνωριστικό στοιχείο συνδέονται. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές αν θα γίνει κάτι τέτοιο ή όχι. Έτσι λοιπόν η κλωνοποίηση ή η τροποποίηση ενός μοναδικού κωδικού είναι σχεδόν αδύνατη και σε Ευρωπαϊκή Ένωση μία λύση χαρτοσύμου θα μπορούσε να είναι καλή επιλογή αρκεί να μην προωθεί τα μονοπόλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα πολύ καλή. Να δώσω το λόγο στον κύριο Λεκένα, γιατί σας έκανε και κάποια ερωτήματα ουσιαστικά, κυρία Μπερτέλ. Τέλο πάντων, ε, θα αναφέρθηκε σε εσά. Ε, πείτε μας και ποιος είστε και τα λοιπά. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και τους δύο προέδρους που με προσκάλεσαν. Είναι μεγάλη χαρά που εκ μέρους της, ε, του συνασυσμού κατά της παράνομης διακίνησης θα ε, κάνω αυτή την παρουσίαση. Η κατάσταση όσον αφορά την δημιουργία ενός, την, κατάσταση της δημιουργίας ενός συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού. Κάνω μια παρομοίαση με την προηγούμενη ομιλήτρια. Μπορεί να είναι με ένα από τα μεγάλα δέντρα του δάσους που τώρα αντιμετωπίζει ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα θα κάνω μια πρώτη παρουσίαση στα γρήγορα και κατόπιν θα απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που μου ζητήθηκε να απαντήσω. Ο λόγος είναι, θέλω να παρουσιάσω τη, για ποιο λόγο έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτή την παρουσίαση που αφορά την παρακολούθηση και τον εντοπισμό, το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού. Αυτά είναι τα ερωτήματα που μου ζητήθηκε να απαντήσω. Εισαγωγικά τώρα, σχετικά με το ποιους δουλεύω. Η Άτος είναι ένας ε, κορυφαίος παίκτη στην ψηφιακή μετατροπή σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ τώρα δοκιμάζουμε την τεχνολογία νομίζω. φτάσαμε. Είμαστε μια εταιρεία περίπου 12 δις ευρώ ε, ε, εσόδων ετησίως. Είμαστε Ευρωπαίος ηγέτης στο χώρο των big data, της παροχής ε, υπηρεσιών clouds και επιχειρηματικές λύσεις και πλατφόρμες. Κάθε χρόνο επεξεργαζόμαστε περίπου 6 δισεκατομμύρια συναλλαγές σε σημεία ε, πωλήσεων, το POS, και επικεντρωνόμαστε στο ένα σκέλος μας, στο παράνομο εμπόριο, την παραποίηση και την φοροαπάτη. Η Atos ε, World Line εν γέννη και το Competence Center πιο συγκεκριμένα ε, έχει δικά, έχει δικά του προϊόντα και λογισμικό. Είμαστε ε, ε, εταιρεία που ενοποιεί συστήματα. Έχουμε δικές μας πλατφόρμες με βάση συγκεκριμένα αιτήματα των πελατών μας από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα. Προσπαθούμε να, να ε, δημιουργήσουμε συγκεκριμένες ειδικέ λύσεις. Σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Μπελέτη, ε, ή έχουμε τεχνολογία όπως το Contentify ή κάποια λύση παρακολούθησης και εντοπισμού και την αξιολογούμε ώστε να δούμε αν είναι κατάλληλη για τους πελάτες μας. Θεωρούμε ότι τα βασικά ε, πλεονεκτήματά μας είναι το, το βιομηχανικό μας DNA. Έχουμε την δυνατότητα να ε, δημιουργήσουμε εξειδικευμένε ηλεκτρονικές λύσεις. Η εμπειρία μα προέρχεται από διάφορους κλάδους, φαρμακευτικά, καπνό, ε, μπύρα, ε, ανταλλακτικά. Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα με την παραποίηση και το παράνομο εμπόριο εντοπίζουμε τις τάσεις της αγοράς και συμμετέχουμε σε διάφορες πρωτοβουλίες όπως η έκθεση 2020 για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό που αν θέλετε μπορώ να σας την ε, επιδώσω. Παρακολουθούμε τις συζητήσεις ε, στο θέμα αυτό επί πολλά χρόνια όπως και την οδηγία για τα φάρμακα. Από το 2014 η οδηγία ε, προϊόντων καπνού προβλέπει ότι το, πρέπει μέχρι το Μάιο του 2019 να έχει υπάρξει ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού. Πρέπει να επισημάνω πόσο πιεστικό είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Βλέπουμε μια χαρακτηριστική ε, ε, ένα χαρακτηριστικό πρόγραμμα υλοποίησης 18 μηνών παρόλα αυτά, επειδή το, το σύστημα δεν, ξέρουμε πώς θα, δεν ξέρει οι παράγοντες πώς θα λειτουργήσει, ε, υπάρχει, ε, υπάρχει δυσκολία. Το θέμα τώρα το, σήμερα. Τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτά τα οποία συζητούνται αφορούν την ε, διατήρηση τακτικής επαφής με όσο δυνατόν περισσότερους εμπλεκόμενους για να γνωρίζουμε τους στόχους. Άρα τα κράτη-μέλη με τα σχετικά υπουργεία και τις υπηρεσίες, αλλά επίσης τους ε, παράγοντες της ε, εφοδιαστικής αλυσίδας οι οποίοι επηρεάζονται, μεγάλους και μικρούς. Επίσης θεωρούμε ότι έχουμε σε επαφή με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ και προσπαθήσαμε να κάνουμε συναντήσεις για να, εκφράσουμε, να ε, παρουσιάσουμε την εμπειρία μας. Αυτό όμως αποδείχτηκε δύσκολο. Επίσης θέλουμε να συμμετέχουμε στις ε, ε, δημόσιες διαβουλεύσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εμπλεκομένων το Μάιο, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ παρα, παρουσίασε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Με βάση αυτά τα οποία μάθαμε από το δίκτυο επαφών μας, αντιλαμβανόμαστε ότι ε, ε συζητώνται οι εξής δυνατότητες το ποιος θα κάνει τι. Η καλύτερη, η προτιμόμενη επιλογή είναι ο, κρατικό, ο κυβερνητικός έλεγχος. Δηλαδή θα, υπάρχουν ε, θα υπάρχει μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο που θα φτάνει μέχρι το σύστημα ε, αποθήκευσης δεδομένων. Θα σκανάρονται από τους διάφορους φορείς μέχρι και τον τελευταίο παράγοντα πριν την λιανική πώληση. Όλοι οι ε, παράγοντες πρέπει να μεταφέρουν τα δεδομένα στο σημείο αποθήκευσης δεδομένων. Ποια είναι η τεχνογνωσία. Παρότι ακούγεται πάρα πολύ τεχνικό, από την κατά την άποψή μας το, ε, το μοντέλο μικτής διακυβέρνησης μοιάζει το πιο λογικό με το να βάζουμε το σύστημα υπό τον έλεγχο των κρατών μελών υπάρχει πλήρης ανεξαρτησία των κατασκευαστών. Δεν ε, αφαιρείται η υποχρέωση από τους ε, παραγωγούς να παρακολουθούν τα προϊόντα τους. Κάποιοι εμπλεκόμενοι με κάθε σεβασμό μπορεί να μην γνωρίζουν τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία. Η πραγματικότητα είναι ότι οποιοδήποτε κώδικας μπορεί να αντιγραφεί από τον οποιονδήποτε. Η ασφάλεια των κωδίκων προέρχεται από μια ανεξάρτητη βάση δεδομένων. Το σύστημα σε αυτή την περίπτωση θα εντόπιζε άμεσα δύο ίδιους κωδικούς. Οπότε θα υπάρχει πρόβλημα και θα ε, ε, συλληφθεί αυτός ο οποίος κάνει την ε, κακή παραγωγή. Τώρα, όσον αφορά το μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων, το συνδυασμένο μοντέλο είναι η προτινόμενη λύση. Κάθε σύστημα αποθήκευσης δεδομένων διαχειρίζεται δεδομένα που έχουν αποκλειστική σχέση, ε, που προέρχονται αποκλειστικά από έναν ε, παραγωγό και υπάρχει ένα σύστημα που δίνει μια ολοκληρωμένη προσε... Ε, από εικόνα όλων των δεδομένων. Ακούμε ότι υπάρχουν ε, αυτοί που προτιμούν το δικό τους σύστημα σε, κάποιο, σε κάποια κράτη-μέλη. Θεωρούμε ότι αυτό οικονομικά δεν είναι συμφέρον γιατί θα έχουμε πολλαπλά αντίγραφα των ίδιων δεδομένων και αυτό απλώς αυξάνει το κόστος το όραμα της Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΤΕ με την προσθήκη αναλυτικών δυνατοτήτων είναι το, η σωστή προσέγγιση. Θα αύξηνε, αύξανε την αποτελεσματικότητα των εθνικών και διεθνών δραστηριοτήτων. Θεωρούμε ότι το σκέλος των analytics θα πρέπει να είναι η λύση για τη μείωση του παράνομου εμπορίου. Θεωρώ ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, οι αρχέ, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, η βιομηχανία και οι αρχές πρέπει να έχουν μια κοινή άποψη. Όσον αφορά τις άλλες ε, προτινόμενες λύσεις, ε, μπορώ να πω απλώς ότι έχουν νόημα και μπορούν να λύσουν το θέμα να ε, βάλουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Υπάρχει μια δυσκολία, το θέμα της νομοθεσίας, γιατί όλα αυτά είναι προς το παρόν ακαδημαϊκές σκέψεις. Έχουμε μαζί, όπως και η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, δύο βασικά ζητήματα που ελπίζουμε ότι θα αντιμετωπιστούν για να είναι επιτυχημένο το σύστημα. Πώς θα εξασφαλίσει η DG Σάντε την συνέχεια του συστήματος, ε, πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια, ε, ένα κεντρικό σύστημα παρακολούθησης που θα λειτουργεί πριν επιτραπεί στους φορείς να αποστείλουν τα ε, προϊόντα. Κάθε σύστημα κάποια στιγμή θα υποστεί βλάβη. Τεχνικά είναι δυνατόν, αλλά δεν βλέπουμε ε, για ποιο λόγο θα υπάρχει αυτό, τι αξία προσφέρει. Δεύτερη πρόβλημα είναι πώς θα εξασφαλίσει η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ ένα λειτουργικό, μοναδικό κωδικό αναγνώρισης. Αυτή είναι μια χωριστή διαδικασία. Όπως είπαμε και στην αρχή, η δημιουργία μοναδικών ε, κωδικών πρέπει να, είναι, να θεωρείται ότι θα προέρχεται από τα κράτη-μέλη. Έρα, σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένου και του καπνού, χρησιμοποιούνται οι οι τυποποιημένοι κωδικοί των κοντέινερ. Και επίσης υπάρχουν οι κωδικοί CC που ε, χρησιμοποιούνται στις παλέτες και, ε, και στα κοντέινερ. Η επιβολή μιας χωριστής διαδικασίας για άλλους κωδικούς θα προκαλέσει πρόβλημα στις υφιστάμενες λειτουργίες. Ενδεχομένως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο και θα δεν θα συμμορφώνονται. Τεχνικά είναι εφικτό. Παρά τα αυτά δεν βλέπουμε ποια είναι η προστιθέμενη αξία παρά μόνον εάν είναι ε, ο στόχος του άρθρου 15 ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων. Τώρα, άλλη ερώτηση. Μπορεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου και εντοπισμού ε, να συνεισφέρει στην επίλυση των, του προβλήματος των παράνομων λευκών, των illicit whites. Θέλουμε να έχουμε πρόσβαση, ε, μια εικόνα της παράνομης παραγωγής αυτών των τσιγάρων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά παράγονται εκτός της Ένωσης με αποκλειστικό σκοπό να εισαχθούν λαθρέα. Σημαίνει αυτό ότι το σύστημα δεν μπορεί να βοηθήσει λοιπόν στο πρόβλημα, την επίλυση του προβλήματο των illicit whites, τα οποία κυρίως προέρχονται από έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι μπορεί να το κάνει. Αν η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος με, με εύκολη συνεργασία με άλλες χώρες ε, εκτός Ένωσης που θα συμμετέχουν και στο πρωτόκολλο FCTC, μπορεί να διευκολυνθεί η κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι κυρίω είμαστε ειδικοί στην τεχνολογία. Δεν είμαστε ειδικοί στο παράνομο εμπόριο. Ποιε είναι οι πιθανότητε οι άλλε χώρε που συμμετέχουν στο πρωτόκολλο FCTC να ε, χρησιμοποιήσουν το σύστημα ελέγχου και εντοπισμού ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπά του. Μόνο αν είναι ανοιχτά τα πρότυπα και εύκολο στη χρήση το σύστημα θα μπορέσουν οι άλλες χώρες να έχουν μια εύκολη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σύστημα που θα είναι εύκολα προσαρμόσιμο με βάση ανοιχτά πρότυπα δεν θα προσφέρει δικαιολογία, τεχνολογική δικαιολογία στις άλλες χώρες. Ένα βαρύ και δύσχριστο τέτοιο σύστημα μπορεί να αποτελέσει αιτία οι χώρες αυτές να απορρίψουν την κύρωση. Έτσι εν κατακλείδη πρέπει να πω ότι αν το μοντέλο που έχει περιγραφεί ε, με, ως την προτινόμενη λύση αποτελέσει τη βάση, όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τον έλεγχο, τη διαλειτουργικότητα, την αναλογικότητα και την αποτελεσματικότητα θα, συμμετέχουν. Στην περίπτωση αυτή, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εντοπισμού και Παρακολούθηση και Εντοπισμού θα μπορέσει να αποτελέσει ε, ε, μια, ένα μέσο για την επίτευξη μιας λύσης όλων όσοι ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση των παράνομων πωλήσεων, κυρίως όσον αφορά ε, τη χρήση των εργαλείων Analytics και Business Intelligence. Σας ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Στρέφομαι σε εσά τώρα αγαπητοί συνάδελφοι να ακούσουμε ερωτήσεις, σχόλια, βέβαια έχοντας υπόψη ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, όλοι θέλουν το λόγο και πρέπει να μπορέσουν να τον πάρουν. Και βέβαια μετά θα πρέπει να έχουν χρόνο και οι προσκεκλημένοι μας να απαντήσουν ή να σχολιάσουν. Έχω λοιπόν ένα κατάλογο ομιλητών ήδη μπροστά μου. Υπάρχει κάποιο που δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα. Μάλιστα, ο κύριο Κον και ο κύριο Αλαφράγκα. Εσά σα έχουμε κύριε. Okay. Uh, so I speaker on my is Ayuso. Η κυρία Αγιούσο είναι η πρώτη και ο καθένας σας θα έχει δύο λεπτά. Κυρία Γιούσου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομη. Όταν συζητήσαμε την οδηγία για τον καπνό, συμφωνήσαμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης. Αυτό όμως δεν μπορούσαν να το κάνουν καπνοβιομηχανίες, αλλά ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Τελικά, στην πράξη, θα γίνει αυτό που προτείνεται από την οδηγία. Δεν είμαι ειδική για αυτά τα θέματα. Αυτό που με ανησυχεί όμως είναι ότι το σύστημα πρέπει να είναι διαλειτουργικό, αποτελεσματικό και να μπορεί να ανταλλάσσει πληροφορίες με τρίτες χώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις εξαγωγές καπνού. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά θα συζητηθούν στο πλαίσιο της δευτερογενούς νομοθεσίας και θα είναι αντικείμενο δευτερογενούς νομοθεσίας. Ποιος αποφασίζει είναι η ερώτησή μου. Ποιε θα είναι οι επιχειρήσει που θα κάνουν αυτή την επιχείρηση χρησιμότητα, παρακολούθηση και έλεγχου. Φαντάζομαι θα είναι αρκετέ. Και τα κράτη-μέλη τι δυνατότητα θα έχουν να λαμβάνουν αποφάσει. Είδατε, δεν έφτασα τα δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγίου Σολή Πρόεδρο. Εξαιρετικό παράδειγμα δώσατε. Ελπίζω να το ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Ο κύριο Παρνιό είναι ο επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Κυρίες Πρόεδροι, καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ που οργανώσατε την ακρόαση αυτή. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί εδώ και κάποια χρόνια είμαι πρόεδρος μιας ομάδας εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς παρεμβαίνουν οι καπνοβιομηχανίες στα πρώτα καπνού. Είμαι δε τακτικό μέλος και στην Επιτροπή Εκτροπής και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ λοιπόν σήμερα το πρωί. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς τους ε, δύο πρώτους ομιλητές, Σεσέλ και Χόφμαν. Τον κύριο Σεσέλ. Πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Από το φύλλο του καπνού μέχρι την πώληση, από το τελικά πρατήρι. Γιατί θέλουμε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο. Και το ερώτημα είναι, θα υιοθετηθεί ένα πλήρες σύστημα που θα επιτρέπει την παρακολούθηση όλης της αλυσίδας παραγωγής μέχρι τα σημεία πώλησης. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή πρέπει πραγματικά να συμμετέχουν οι καταναλωτές, θα πρέπει να υπάρχουν εμφανή αρτιστικά ασφαλείας για να μπορεί κανείς να τα διαβάζει, παρουσιάρει με τα smartphone, για να καταλαβαίνει αυτό μας που πρόκειται. Αυτό του είδους η χνηλασιμότητα είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να δώσει περισσότερη εξουσία και περισσότερες πληροφορίες στους καταναλωτές. Συμφωνείτε μαζί μου. Και έρχομαι στην κυρία Χόφμαν. Όταν θα έχουμε σε επίπεδο ένωσης ε, την εχνηλασιμότητα, την ανεξάρτηση, όπως αποφασίσαμε το 20 Μαΐου 2019, οι τρεις συμφωνίες συνεργασίας που έχουμε με, Japan Tobacco International και Imperial Tobacco έχει νόημα να συγχυστούν. Japan Tobacco λύγει το 2022. British Tobacco και Imperial Tobacco λύγουν το 2030. Όταν θα έχουμε όμως συνολικά αυτή την χνηλασιμότητα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε αυτούς τους διακανονισμούς τους φιλικούς του 2004 μεταξύ Philip Morris International, που δεν την έχουμε, τα την είχαμε και με την Κομισιό, διότι μας επέτρεπε τότε να έχουμε αυτή την παρακολουθία και τον εντοπισμό με πρωτοβουλία των επιχειρήσεων. Τώρα όμως προσανατολιζόμαστε, είναι σαφές, προς έναν άλλο στόχο και τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ για την εφαρμογή των άρθρων 15 και 6 οδηγία, 15 και 16. Ε, για τα πρώτα. Φυσικά και είναι σημαντικό το σύστημα παρακολούθησης ε, και εντοπισμού να είναι ανεξάρτητο, το λένε όλοι. Το σύστημα λοιπόν παραγωγής κωδίκων και εκτύπωσης αυτών θα πρέπει να μην μπορεί να παραβιαστεί και να ελέγχεται από τις εθνικές τελωνιακέ αρχές. Άρα η Κομισιόν θα πρέπει να φροντίσει εξωτερικοί ελεγκτές που θα επιφορτιστούν με τον έλεγχο της βάσης δεδομένων είναι εξάρτητοι. Αυτό σημαίνει και ότι το σύστημα που θα δημιουργήσουμε θα πρέπει να σέβεται επακριβώς τις διατάξεις του ε, πρωτοκόλου του ΠΟΗ για το λαθρεμπόριο πρώτων καπνών. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα που θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει εμπρόθεσμα μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει η οδηγία. Θέλουμε να είναι επιχειρησιακό, λειτουργικό, να μην είναι περιττό, να υπάρχουν ε, δυνατότητες ε, αλληλεπίδευσης με τα ανοιχτά συστήματα. Δεν συμφωνώ με αυτούς που θέλουν να μας ε, κλείσουν σε μια παγίδα ενός αφηγήματο που λέει ότι από τη μία έχουμε τις καπνοβιομηχανίες και από την άλλη την ενιαία λύση που είναι στα χέρια ενός και μόνου παράγοντα φορέα εκμετάλλευση. Υπάρχουν ε, τεράστια προκλήσει και συμφέροντα. Εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω. Υπάρχουν και πάρα πολλέ ΜΜΕ. Έχω και προς τους ε, προσκεκλημένους μας μια ερώτηση. Το κόστος των διαφόρων σεναρίων που εξετάζει η Κομισιόν, ποιο είναι, ποιος θα το αναλάβει το κόστος, οι εθνικές αρχές, η καπνοπαραγωγή, ο ιδίο κτλ. και ανάλογη. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Αγκροστέτ, επόμενο ομιλητή. ο κύριο Χολβένη. Χολβένη. Εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πω όμως τη γλώσσα μου, αν μου επιτρέπετε. Ως μέλος της Επιτροπής ΕΝΒΗ, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ευρύτερα την εικόνα. Περί τίνος πρόκειται εδώ. Άκουσα τις τρεις παρουσιάσεις με πολύ ενδιαφέρον. Έχω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Πρώτον, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ό,τι και αν κάνουμε το κάψιμο ποτέ δεν θα είναι υγιεινό. Και όσο και αν μιλάμε για δουλειές και για έσοδα από τη φορολόγηση του καπνού. υπάρχει το θέμα της υγείας. Το επόμενο. Πώς μπορεί η Κομισιόν να εξασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα σύστημα που δεν θα ε, μόνο τους μεγάλους και θα εκτοπίσει τους μικρούς, γιατί μιλάμε για χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τι θα συμβεί επίσης χώρες που είναι εκτός Ένωσης. Αυτά τα παράνομα λευκά έρχονται κυρίως από Ουκρανία, Ρωσία, Λευκορωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα κάνουμε γι' αυτό. Όπως και η κυρία Γκροστέτ, τι θα γίνει με τους μικρούς ε, παραγωγούς καπνού. Δεν θα πρέπει κάπως να περιοριστεί το βάρος που φέρουν. Όσον δε αφορά το πρωτόκολλο του ΠΟΗ, προβλέπονται πέντε χρόνια για τον ετοπισμό. Εμείς όμως έχουμε ένα χρόνο μέχρι το 2019. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να δοθεί περισσότερο χρόνο στους μικρούς παραγωγούς για να προετοιμαστούν, για να μην τους καταστρέψουμε και να μην χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κύριε Μπον, ε, τα ερωτήματά μου έχουν να κάνουν με το CODENTIFY Είπε η Κομισιόν επίσης και για τα εννέα γνωστικά στοιχεία, ότι αυτά είναι ανεξάρτητο τρίτο μέρος θα τα παράγει. Τι θα πει αυτό ανεξάρτητος τρίτος, ποιος θα είναι αυτός. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 15, 8, ελεγκτής, πώς θα ξέρουμε ότι θα είναι ανεξάρτητος, αν οι τέσσερι, ε, έχοντας υπόψη μας ότι οι πελάτες ε, των τεσσάρων μεγάλων ελεγκτών ε, μεταξύ των πελατών στο υπάρχουν και καπνοβιομηχανίες. Ό,τι αφορά την ε, ειδική ομάδα για το λαθρεμπόριο, ποιοι περιλαμβάνονται. Μόνο τα κράτη-μέλη αναφέρονται στο ίντερνετ. Ορίστηκαν από τα κράτη-μέλη, ανεξάρτητοι πράγματι αυτοί οι άνθρωποι. Ποιοι είναι. Ούτε όλα μου είχε απαντήσει. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, θα ήθελα να ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σάνι. Εσείς, ναι, εσείς, ο κύριος Σάνι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τις παρουσιάσεις πολύ προσεκτικά. Και από τη στιγμή που ήρθα στην αίθουσα ε, μέχρι τώρα αυξήθηκαν οι ανησυχίες μου κατάλαβα ότι δηλαδή υπάρχουν κάποιες προθεσμίες που πλησιάσουν στο τέλος τους. Και πρέπει να συμφωνήσω με τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένως και εξέφρασε ανησυχία για την προθεσμία το 2019. Είναι πάρα πολύ κοντά. Γι' αυτό ρωτώ την Κομισιόν πότε σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διεπηρεσιακές διαβουλεύσεις και να ξεκινήσει η δημοσία διαβούλευση για την σχέδιο εφαρμοστικής πράξης. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι ότι η καπνοβιομηχανία και ιδίω οι μικρότεροι οι διανομείς δεν θα μπορούν να σεβαστούν την νομοθεσία μέχρι την ημερομηνία αυτή. και θέλω να αναφερθώ σε κάτι που είπε εκπρόσωπος της Κομισιόν. Είπα ότι έκαναν διαβούλευση με τη βιομηχανία και με τους εμπόρους. Μόνο όταν ήταν απολύτως απαραίτητο. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ε, στους παίκτες της αγοράς. Um, ε, ε, Διαφορετικά, θα κινδυνεύουμε να καταρρεύσει το όλο σύστημα. Και φυσικά δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους ομιλητές ε, για τους παρουσιάσεις τους. Έχω τρεις ερωτήσεις. Η μία αναφέρεται σε αυτά που είπε και ο κ. Μπολέν μόλις τώρα, αναφερθήκατε στο άρθρο 15, το οποίο θεσπίζει ένα ανεξάρτητο σύστημα εχνηλασιμότητας και εντοπισμού και στην οδηγία για τα προϊόντα καπνού. Στο άρθρο 15 αναφέρεται ότι οι κατασκευαστές πρέπει να διαλέξουν έναν ανεξάρτητο φορέα για την αποθήκευση των δεδομένων, πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτοί οι ανεξάρτητοι ελεγκτές και συνεργάτες όντως είναι ανεξάρτητοι και θεωρούνται ανεξάρτητοι. Ποια κριτήρια υπάρχουν για να το απαντήσετε αυτό. Κάποια στιγμή η κυρία Λορένς Περτελέτη είπε ότι δεν ε, είναι ε, δυνατόν να βρούμε σε ποιο σημείο στην ελισίδη εφοδιασμού τα νόμιμα παρασκευασμένα προϊόντα έχουν διοχετευτεί στην παράνομη αγορά. Υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό που δείχνει ότι η παράνομη αγορά είναι αποτελείται ουσιαστικά από ε, γνήσια προϊόντα καπνού και όχι από παραπημένα ε, προϊόντα ή από φτηνά λευκά. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για το αν έχει σχεδιαστεί το σύστημα εχνηλασιμότητας και εντοπισμού για να ελέγξει αυτή την παράνομη αγορά γνήσιων τσιγάρων και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ε, μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει και μας δείχνουν οι στατιστικές. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μαζερόνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και ενημέρωση. Έχω κάποιες ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κυρία της Όλαφ. Τι μέτρα έχει λάβει η Κομισιόν για να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση θα δημιουργήσει φραγμούς στις εξαγωγές προϊόντων καπνού τα οποία παρασκευάζονται στα κράτη-μέλη της Ένωσης έχετε έρθει σε επαφή ε, με τους εταίρους ή ε, πως υπάρχουν άλλα καθεστώτα τα οποία έχουν να κάνουν με τα προοριζόμενα για εξαγωγή προϊόντα. Δεύτερο ερώτημα, πώς θα εξασφαλίσετε ότι το ευρωπαϊκό σύστημα είναι συμβατό με τα άλλα συστήματα που υπάρχουν σε παγκόσμιο και τρίτον. Αληθεύει ότι η Κομισιόν προτείνει να δημιουργηθεί ένα οργανισμός ευρωπαϊκός που θα αναλαμβάνει τα σχετικά τα στον τομέα των προϊόντων καπνού. Τι αρμοδιότητες θα έχει αυτός ο νέος οργανισμός. Ευχαριστούμε κύριε Μαζουρόνη. Σε κυρία Γκαρτίνη. Κυρία Γκαρτίνη, ευχαριστώ. Λοιπόν, να περνώ κατευθείαν στις ερωτήσεις, γιατί συμφωνώ με όσα είπαν οι συνάδελφοι η και Κρουστέτ. Είπαν πολλά με τα οποία συμφωνώ. Και εγώ βλέπω πολύ αισιόδοξη την προσέγγιση της Κομισιόν που είπε ότι μπορούμε να σεβαστούμε τις προθεσμίες. Εγώ νομίζω ότι είναι μεθαύριο αυτό και μου δημιουργεί κάποια ανησυχία για το ποιο μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα σε σχέση με τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα ενός συστήματος που θα έχει γίνει τόσο γρήγορα σε ποια πραγματικά στοιχεία βασίζεται την αισιοδοξία σας και κατόπιν ανησυχώ πάρα πολύ για αυτό το σύστημα ιχνηλασιμότητας που θα μπορούσε ουσιαστικά να πάρει την μορφή μονοπωλίου. Εγώ νομίζω ότι το μονοπόλιο καταφέρεται των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως κατά του ελεύθερου ανταγωνισμού και της ελεύθερης συμμετοχής της υπηρεσίας. Εμείς χρειαζόμαστε συστήματα εχνηλασιμότητας που να βασίζονται οπωσδήποτε σε ανοιχτά πρότυπα και φυσικά με λογικό κόστος και για τους μικρούς οικονομικούς φορείς. Εγώ νομίζω ότι στα σημεία αυτά θα πρέπει να είμαστε κάθετοι. Και αν δεν πράξουμε έτσι, σκεφτόμαστε κατά τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ βλέπω ότι πιο ενδιαφέρουσα συνεισφορά σε σχέση με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου γίνεται από του τελωνιακού. Μίλησε η Κομισιόν με του τελωνιακού που έχουν εμπειρία στο θέμα αυτό και μπορεί να έχουν ιδέε και πολύ συγκεκριμένε συνεισφορέ ε, να κάνουν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Το κύριο Ähm, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πριν έρθω εδώ στο ε, Κοινοβούλιο, ασχολούμουν με θέματα εφορίας ε, και έλεγχα, εφορολογικές δηλώσεις, άρα ξέρω λίγο πολύ για απάτες. Ε, ε, σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, την επιτάχυνση των διαδικασιών στα κράτη-μέλη και όλα τα σχετικά πραγματικά είναι σημαντικά και πρέπει να, πλησι... να συμπληρώσουμε με αυτόν τον τρόπο το σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης. Ε, σε ό,τι αφορά τις προθεσμίες ε, στο Συμβουλίο Υγείας υπήρξαν αντιδράσεις από διάφορα κράτη-μέλη. Άρα πώς πράγματι πιστεύετε ότι θα τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες ε, και τι θα γίνει με αυτές τις ε, διαδικασίες ε, που θα πρέπει, αν ισχύσει αυτή η προθεσμία του 2019, τι θα γίνει με τα ευαίσθητα προϊόντα. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν καπνίζω εγώ. Παρ' όλα αυτά με ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση πάρα πολύ και όπως και άλλοι συνάδελφοι θέλω να εστιάσουμε στις προθεσμίες. Δηλαδή αν αυτά τα μέτρα, τα εφαρμοστικά, θέλετε να εφαρμόζονται για, από το 2019 για τον καπνό και για τα υπόλοιπα από το 2025 και μετά, ενδιαφέρον είναι να δούμε τι σχεδιάζει η Κομισιόν. Και πρέπει εμείς ε, ως κοινοβούλιο ε, να δούμε τι έχουμε να κάνουμε. Γιατί αν θέλουμε ε, να τηρηθούν οι προθεσμίες πρέπει να έχουμε αντιδράσει μέχρι το τέλος του έτους. Σίγουρα διαλειτουργικότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα είναι η λέξη κλειδιά και σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει αντιμονοπολιακό αποτέλεσμα, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να θέσει διεθνή πρότυπα. Αυτός είναι ο ρόλος μας που θα μπορούν να τα μιμηθούν άλλες περιφέρειες δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα πολύπλοκο σύστημα ή υπερβολικά δαπανηρό, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που θα προσφέρει επιλογές και θα μπορεί να υιοθετηθεί και από άλλες περιοχέ του κόσμου. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε πώ θα επηρεαστεί η απασχόληση. Δεν ξέρω αν το σκέφτεται αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ επίση και το γεγονό ε, το κατά πόσο εξετάζεται να εφαρμοστεί κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα επειδή για κάποια από τα προϊόντα πάρα πολύ σύντομα, λίγη προθεσμία και θα πρέπει να εφαρμοστούν. Και ήθελα να μου πείτε, ε, σε σχέση με αυτό που η κυρία Γκραντίνη, και τι άποψη έχουν τελειώσει για το παράνομο εμπόριο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζόμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ φυσικά συμφωνώ ε, σε σχέση με αυτά που είπε ο προλαλής σας. Μέχρι τα τέλη του χρόνου σίγουρα εμείς θα πρέπει να δούμε την εκτελεστική πράξη με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Ε, τελικά τι κάνει η Κομισιόν, μας πιέζει απλά και μόνο για να πετύχει να τηρηθούν οι προθεσμίες. Δεν υπάρχει τότε επιμήκυνσης, ίσως να υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος. Δεν, δεν ξέρω, δεν, δεν το βλέπω εγώ να μπορούν να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να το θέσω, αν μπορεί να αλλάξει. Σε ό,τι αυτά τα διεθνή πρότυπα, το είπε και ο κύριος Αλαφράγκα, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά υπάρχουν συστήματα εντοπισμού ε, ήδη στην ε, αγορά, όπως για τα ψάρια για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί η Κομισιόν λοιπόν. Έχει μελετήσει αυτά τα συστήματα, έχει υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές. ξέρω γιατί γελάτε. Ε, γιατί γελάτε για τα ψάρια, για τον καμποτέσπα. Ε, και έπειτα σε, αυτό, σε σχέση με αυτό το νέο σύστημα εντοπισμού και παρακολούθησης ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δομές που υπάρχουν, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέες. Σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά προγράμματα των κρατών μελών ε, ε, σκέφτεται να τα αξιοποιήσει, έχει λάβει υπόψη τις εμπειρίες. Και τέλος, ό,τι αφορά έναν ορισμό για τα πρώτα καπνού. Από τον παραγωγό μέχρι τον τελευταίο που συμμετέχει στην αλυσίδα μέχρι το σημείο πώλησης. Όλοι αυτοί θεωρούνται ότι συμμετέχουν. Σημείο πώλησης είναι το σημείο ε, διάθεση των προϊόντων στον καταναλωτή. Αυτό λέει η οδηγία. Αλλά υπάρχουν πολλοί λιανοπολιτές που χρησιμοποιούν κεντρικέ αποθήκες και υπάρχουν και θηγατρικέ. Αλλά πολλές φορές, ε, μάλλον αυτές οι ιδιωτέ αποκλείονται ως ε, σημείο πρόκληση και υπάρχει σύγχυση με αυτό το θέμα. Τι είναι αυτά τα σημεία τελικά, ποια είναι, θα μπορούσε να τα ξεκαθαρίσει αυτή η Κομισιόν. Αυτή σε αποθήκες τελικά προμηθεύονται οι λιανοπολιτές. Εμπίπτουν, δεν εμπίπτουν, είναι πολύ... Η κυρία Κάντεμπαχ, ευχαριστώ. Πολύ σύντομο ερώτημα. Εμπειρίες, αν υπάρχουν, με το σύστημα αντιμετωπισμού και παρακολούθησης. Σε ό,τι αφορά τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, για τα ψάρια δεν, το, δεν μπορώ να το καταλάβω, ούτε που το φαντάζομαι. Ε, για τα φάρμακα όμως, μήπως έχετε δει αντίσταση. συστήματα. Κυρία Γκρέσλη, θα σας δώσω τώρα σε εσά το λόγο και μετά θα σας δώσω και την παιδρία. Ευχαριστώ πολύ. Στον κύριο Σεσέλ, είχα κάπως απογοητευτεί από την αρχή σας παρουσίαση, περιμέναμε κάτι παραπάνω για το τι σκέφτεστε, τι προβλέπετε. Είναι σημαντικό για εμάς. Γιατί αν δεν προσέξουμε, κάθε μικρό σημείο πώλησης, ε, ταμπά, ε, κιόσκ, ε, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πάρα πολύ πολύπλοκο σύστημα και αυτό πρέπει να το προσέξουμε με αυτό το σύστημα το οποίο έχετε σκεφτεί, ε, θέλετε να είναι ένα ε, επιχειρησιακό και ανοιχτό σύστημα. Πού, πόσο έχετε προχωρήσει, έχετε έρθει σε επαφή επίσης με τη γραμματεία του FCTC. Γιατί σίγουρα πρέπει ό,τι κάνουμε εμείς να είναι συμβατό με το FCTC. Και για την όλα μια ερώτηση. Εσείς συμμετέχετε σε αυτές τις συζητήσεις, στον προβληματισμό για το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού και στο πώς ακριβώς ε, θα οργανωθεί το όλο σύστημα. Είπατε 3,8 εκατομμύρια τσιγάρ τσιγάρου 2010 και μετά. Από αυτά πόσα ήταν πρωτότυπα, ε, αυθεντικά προϊόντα. Παρακαλώ να απαντήσετε σιγά σιγά. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να ενδεχομένω να απαντήσω στο σημαντικό ζήτημα του χρόνου. Το γνωρίζει απολύτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπα πριν, στόχος μας είναι και είμαστε εντός προγράμματος, προβλέπουμε την ε, υιοθέτηση των νομοθετικών πράξεων μέχρι το τέλος του χρόνου. Πράγμα που πιστεύουν θα επιτρέψει επαρκή χρόνο για την εφαρμογή τους. Σύμφωνα με τους κανόνες της ε, καλύτερης, ε, του better regulation, έχουμε ε, ε, σκοπό να, στο τέλος του καλοκαιριού να ενημερώσουμε πριν από τη θέσπιση. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία του 2019 ισχύει για τσιγάρα και για τσιγάρα που τα στρίβει κανείς μόνος του. για τα υπόλοιπα είναι ο Μάιος του 2024. Το άλλο θέμα είναι το κρίσιμο ζήτημα της ανεξαρτησίας πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κριτήρια είναι σαφή και κοινά για την επιλογή και την έγκριση των ανεξάρτητων τρίτων. Ανεξάρτητος σημαίνει ανεξάρτητος από την καπνοβιομηχανία, φυσικά σύμφωνα με το πρωτόκολλο FCTC. Για τον λόγο αυτό σκοπεύουμε να συμπεριλάβουμε μια σειρά από βασικά κριτήρια στο σχέδιο νομοθετήματος που συζητώνται ακόμα με τα κράτη-μέλη. Είναι πιθανόν να επικεντρωθούν σε μια σειρά στοιχείων όπως αξιολόγηση της ανεξαρτησίας των φορέων από την καπνοβιομηχανία, οικονομικά, διοικητικά και επίσης την, ε, ε, την, να υπάρχουν δηλαδή προστατευτικά τείχη που να είναι αποτελεσματικά, τα firewalls. Και θα πρέπει επίσης να στηριχθούν διάφορα πρότυπα στην αξιολόγηση ανεξαρτησίας. Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το κόστος που ετέθη. Προσέξαμε πολύ το θέμα αυτό στην μελέτη επιπτώσεων και στην διατύπωση των προτάσεών μας. Ε, καταρχήν, να σας διαβεβαιώσω ότι οι λιανοπολιτές. Φυσικά δεν υπάρχουν βασικές απαιτήσει που να προβλέπονται από αυτούς, πέρα ενδεχομένως από μια καταχώρηση εγγραφή σε ένα μητρό ε, λιανικού εμπορίου. Πιστεύω ότι αυτοί θα είναι οι νόμιμοι πολιτές που θέλουν να αποφύγουν τον αθέμητο ανταγωνισμό από του παρανόμου. Το κόστος έχει επίσης ληφθεί υπόψη σοβαρά και μπορώ να σα πω ότι καταδείξαμε σαφώς ότι το κόστος ε, αναμονάδα σε πακέτο, αναπακέτο θα είναι ελάχιστο αν όχι αμεληταίο. Η αποτελεσματικότητα δηλαδή όσον αφορά το κόστος του μέτρου είναι πολύ υψηλή. Τώρα, το θέμα των τρίτων χωρών και αυτό είναι ένα ζήτημα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες ολόκληρο τον κόσμο θα εφαρμόσουν, καταρχήν θα υιοθετήσουν, θα κυρώσουν και θα εφαρμόσουν το πρωτόκολλο. Είναι κρίσιμο αυτό γιατί είναι η μοναδική ελπίδα που υπάρχει παγκοσμίω να υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου. Θεωρούμε ότι αν κινηθούμε γρήγορα είμαστε ε, ε, ισχυροί και δείξουμε πώς μπορεί να γίνει, θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε τις τρίτες χώρες να θεσπίσουν ε, παρόμοια ή συμβατά έστω μέτρα. Το θέμα είναι η Γραμματεία της FCTC ε, με την οποία συνεργαζόμαστε. Καταρχήν θέλουμε ό,τι κάνουμε να, είναι, να ευθυγραμμίζεται πλήρω με τις διατάξεις του πρωτοκόλου και να μπορούν να το ε, θεσπίσουν και άλλες χώρες. Είναι σημαντικό να κινηθούμε το ταχύτερο δυνατόν γιατί αυτό πιστεύω θα βοηθήσει να επιληθούν μια σειρά από τεχνικά ζητήματα για τα οποία ρωτούν οι τρίτες χώρες. Όπως ήδη επισημάνθηκε το πεδίο ε, του συστήματος είναι να εντοπιστεί η στιγμή και το σημείο ε, που το προϊόν ξεφεύγει από την νόμιμη οδό και μπαίνει στην παράνομη. Τα δεδομένα που θα διατίθενται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς σκοπούς. Το συζητάμε με τα κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα μπορώ να δώσω. Τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση πιο εύκολα να εντοπίσουν ευνίδιες αλλαγές. Παραδείγματος χάρη, κάτι που γίνεται σε επίπεδο ε, λιανικού εμπορίου και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Δηλαδή μια μορφή που αλλάζει ξαφνικά. Σήμερα, σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Το σύστημα θα το επιτρέπει. Θα αποτελέσει αυτό αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ε, δολιοφθοράς ή της, ε, ε, των παράνομων λευκών. Επίσης θέλουμε να εμπλέκονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι Μα ενδιαφέρουν οι, κυρίως η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 3 του FCTC που ε, αναφέρεται στην, ε, ε στις επαφές ε, του καπνοβιομηχανίας και τους, ε, τους νομοθέτες αλλά βεβαίως δεν σημαίνει ότι η καπνοβιομηχανία δεν μπορεί να δώσει την άποψή της. Η διαδικασία ήταν ανοιχτή και διαφανής. Όλοι μπορούν να το πούν αυτόν. Είμαστε σε στενή επαφή κυρίως με τις διοκτικές αρχές γιατί φυσικά πρέπει να σχεδιάσουμε ένα σύστημα σύστημα που κυρίως αυτούς θα διευκολύνει και πήραμε πολύ χρήσιμες πληροφορίες από τελωνιακούς και, άλλους, ε, ε, και, αρχέ. και άλλες διοκτικές αρχές. Οι επαφέ συνεχίζονται. Νομίζω ότι απάντησε σε όλε τι ερωτήσει. Αν κάτι παρέλειψα, παρακαλώ μου το πείτε. Χόφμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μου ετέθησαν και εμένα κάποια ερωτήματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσω, αλλά θα, θα τα πω αγγλικά παρόλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Σπανιό νομίζω με ρώτησε για τις τρεις συμφωνίες ε, για τον καπνό κατά πόσο είναι ανάγκη να συνεχιστούν αυτές οι συμφωνίες με την καπνοβιομηχανία εφόσον θα έχουμε πλέον το σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού στο πλαίσιο τη οδηγία ε, για τα πόντα καπνού. Πολύ σωστά είπατε κύριε Πανιό ότι έχουμε αυτές τις τρει συμφωνίε. Όχι η Κομισιόν όμως είναι συμβαλλόμενο μέρο. σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη. Είναι συμβαλλόμενο μέρο. Το 2022 λήγουν οι συμφωνίες. Και το 2030. Σε ό,τι αφορά, επαναλαμβάνω και είναι τέλειο, το σύστημα παγκοσυντοπισμού. Αν δούμε μόνο τον του καπνού, περιοριζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο σύστημα, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό το πρωτόκολλο FCTC του ΠΟΗ, το επικαμάρτες ΕΣΕΛ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο στην Ένωση παρακολούθηση και τοπισμός δεν βοηθάει να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο στα σύνορα. Χρειάζεται το πρωτόκολλο ευσύτηση. Αλλά δεν ισχύει ακόμη. Πέντε χρόνια υπάρχει μεταβατική περίοδος, άρα θα χρειαστεί χρόνος. αλλά το ε, πεδίο εφαρμογή, η εμβέλεια, αν θέλετε, των συμφωνιών με τι ταπεμπικά είναι παγκόσμιο ισχύουν στο παγκόσμια κλίμακα. Αυτό που είναι όμως πιο σημαντικό ακόμη είναι ότι αυτές οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και κάποιες άλλες διατάξεις για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος, για τη δέωση επιμέλεια και το καθεξής. Άρα υπερβαίνουν το πεδίο πολύ εντοπισμό. Το τελευταίο που θέλω να προσθέσω σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι όλες οι συμφωνίες περιλαμβάνουν μια ρήτρα που λέει ότι υπερτερεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει οι παρασκευαστές καπνού πάντοτε να συμμορφούνται προς τις ε, νοσιακές διατάξεις και τις διεθνείς. Δεύτερη ερώτηση ήταν, που είναι η ερώτηση, α, ναι, αρκετοί βουλευτές ανέφεραν τα τελωνία και σε ποιο βαθμό συμμετέχουν σε συζήτηση. Συμμετέχουν οι τελωνικές αρχές στο σχηματισμούς του Συμβουλίου του Σχετικούς. Πριν από δέκα μέρες είχαμε μια συνάντηση το, με τους Γενικούς Διευθυντές Τελωνίων ε, σε σχηματισμό του Συμβουλίου που συστήθηκε αυτό το θέμα. Ο αρμόδιος τα Σαντέ και εγώ ήμουν εκεί και απαντήσαμε σε ερωτήσει. Άρα υπάρχει διάλογος και με τα τελωνία. Ένα άλλο ερώτημα ήταν να πω κάποιον άλλο και αφορούσε την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Και είπε ότι ήταν η κυρία εκεί, Είπε ότι δεν αναφέρει τα ονόματά τους ή όλα. Εμείς είμαστε διαφανείς, κυρία μου. Έχουμε αυτή την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο από την και εκεί συμμετέχουν εμπειρογνώμες από τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει κανένα ιδιωτικό συμφέρον. Είναι μια συνάντηση με εμπειρογνώμονες από τον κλάδο, οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία ορίζουν αυτούς που στέλνουν εκεί και αυτό μπορεί να αλλάξει. Τα κράτη-μέλη δεν είμαστε εμείς αυτοί που αποφασίζουμε. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Γκρέσλα. Τα 3,8 δις τσιγάρων που είπα και εγώ στην αρχή. Τα έχετε τα στοιχεία και ε, στην έκθεση του Μαΐου 2017. Με βάση τα κράτη-μέλη, τα στοιχεία από το 2013 Έξι από τις, πιο, έξι από τις δέκα ε, μεγαλύτερες κατασκευές ποσότητες αφορούσαν λευκά ε, σιγά Εμείς διευκολύναμε τη διαδικασία ε, ένα δις περίπου και τα τελευταία χρόνια το 9% ήταν φθηνά λευκά. Αυτά είναι τα στοιχεία μας. Άρα παραμένει το πρόβλημα με τα φθηνά λευκά και μάλιστα επιδεινώνεται. Το τελευταίο. Είπατε αν συμμετέχουμε στη συζήτηση για την παρακολουθήση και τον Η γάμα δέλτα σαντέ είναι η κύριοι του εγχειρήματο, ε, οι άρχοντες της, όχι του διαστήματος, αλλά αυτής της συγκεκριμένης ε, διαδικασίας. Και συμμετέχουμε εμείς, όπως είχαμε τα τάξουτ, Συμμετέχουμε δηλαδή σε διπηρεσιακές συναντήσεις και ελπίζουμε και να συμμετέχουμε και στις, κατε... στις αγραμμοστικές πράξεις, ε, στις συναντήσει αυτές συναντήσεις, στις εκτελεστικές πράξεις. Μαζί με τη γόμα ΣΑΝΤΕ και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ υπογραμμίζετε πολύ σωστά πόσο σημαντική είναι η διεθνή πτυχή. Κύριε Καρντίνη λέει ότι δεν απαντήσατε το ερώτημά της για τα μονοπόλια. Μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Αν με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποτρέψουμε, να αποφύγουμε τα μονοπόλια. Ναι, αυτή είναι η πρόθεσή μας. Η πρόθεσή μας είναι να θέσουμε τα κριτήρια και να επιτρέψουμε να υπάρχει ανταγωνισμό στην εφαρμογή των κριτηρίων. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ναι η απάντηση στην ερώτησή σας, θα το διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπερτελέτη, το έχει το λόγο. actually not... Δεν, ε, I will... είμαι σίγουρη αν απευθύνθηκε κάποια ερώτηση προς εμένα για να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Πολλοί βουλευτέ έκαναν σχόλια για την προθεσμία. Αυτό με εντυπωσίασε. Και ενώ νομίζω ότι είναι σημαντική η προθεσμία, νομίζω ότι αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι είναι καλό το σύστημα, ότι είναι στεγανό απέναντι στην καπνοβιομηχανία και ακόμη και αν καθυστερήσει λίγο θα ήταν αυτό το τέλος του κόσμου δεδομένου ότι αυτό το σύστημα που οικοδομούμε θα είναι το παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή την ανησυχία για την προθεσμία. Γιατί γίνεται τόσο, ε, τόσο φασαρία γι' αυτό. Ευχαριστώ για τη χαλαρότητα γενικώ που δείξατε, ο κύριος Λεκέ. Ευχαριστώ να δηλώσω ότι ως ένα παρόχος ε, τεχνικής υπηρεσίας ε, εξακολουθώ να είμαι συνεπαρμένος. Πρόκειται για ένα ε, σύστημα πρωτοπόρο που θα εφαρμοστεί ε, για τους καταναλωτές ε, θα επικεντρωθεί στο να εντοπίσει τις απειλές, τουλάχιστον έτσι βλέπουμε εμείς τα πράγματα και θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουν καλύτερα. Θα έχουμε ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε το παράνομα εμπόριο. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να καταπολεμήσει όλους τους πιθανούς τρόπους λαθρεμπορίου, γιατί διαφορετικά θα έχουμε ένα σύστημα που δεν θα δουλεύει. Έτσι λοιπόν ε, οι εταιρείε ε, IT συνήθως ε, έτσι διαχειρίζονται τα προϊόντα τους με τους πελάτες τους. Ελπίζω να σας βοήθησα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή στη συζήτηση. Ευχαριστώ και την κυρία Γκρέσλε για την ανάληψη της πρωτοβουλίας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα και είναι και αναγκαίο και νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε το χρόνο για να αναπτύξουμε ένα σύστημα αξιόπιστο και μοντέλο όπως είπατε για τον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Παρακαλώ να παραμείνετε και για την επόμενη ανταλλαγή απόψεων. Θέλω να ευχαριστήσω στα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, και τους ε, προσκεκλημένους. Θέλω να προχωρήσουμε, γιατί εμείς έχουμε εδώ από την Επιτροπή του Προπολογισμού να δούμε ένα ακόμη θέμα που είναι η ειδική έκθεση 33 του 2016 η ειδική έκταση για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η γήτρια είναι η συνάδελφο Κάντεμπαχ. Και από το Ελληνικό Συνέδριο με τον κύριο Βέσπερκ, που θα πάρει το λόγο ευθύ αμέσω για να μας παρουσιάσει. Έχουμε 10 λεπτά παραπάνω από τις 12.30. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα. Έχετε το λόγο κύριε Βέσπεργκ. Please, Mr. Vesberg, you have the floor. Κύριε το λόγο. Okay, I ε, ε, ε, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει θα πάρω το λόγο, έχω τη χαρά να σας στείλω είχα τη χαρά να στείλω την ειδική έκθεση για τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης και το πώς υπάρχει, λειτουργήσει η ανταπόκριση σε καταστροφές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λίγο ενοχλητικά όλα αυτά. Μήπως μπορούν Παρακαλώ καθίστε, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ καθίστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Παρουσιάσαμε από κοινού την έκθεση αυτή ε, στον Ιανουάριο του 2017 με τον Επίτροπο κ. Στυλιανίδη. Με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι κλεισμένα σε ένα εργαστήριο αλλά ε, συνεργάζονται για να είναι αποδοτικά. Οι πολιτικές της Ένωσης, ε, ε, γιατί είναι αποδοτικές οι πολιτικές της Ένωσης και ταυτόχρονα να διαφυλάζονται τα συμφέροντα των πολιτών. Όσον αφορά η καταστροφή μπορεί να χτυπήσει ανα πάσα στιγμή οπουδήποτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί ε, είτε σε ανθρωπογενείς είτε σε φυσικές καταστροφές αλλά οι οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να είναι σοβαρές. Πρέπει να ε, να μελετηθεί η απόδοση των κονδυλίων για να δούμε πώς μπορεί το εκτελεστικό της σκέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, να ε, προγραμματίσει πραγματικά μελετήσαμε το συντονισμό των, ε, της ανταπόκρισης σε καταστροφές εκτός της Ένωσης από το 2014 που συστήθηκε αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας. Περιλαμβάνει τη διευκόλυνση του συντονισμού με συμμετέχοντα κράτη, άλλα θεσμικά όργανα και φορείς, τα Ηνωμένα Έθνη, της, την πληγήσα χώρα και άλλους ε, παράγοντες ως ε, μέλος υπεύθυνο για την έκθεση αυτή θέλω να σας στείλω το βασικό μήνυμα. Δηλαδή η Επιτροπή σε γενικές γραμμές ήταν αποτελεσματική στη διευκόλυνση του συντονισμού των, της ανταπόκρισης σε καταστροφές εκτός της Ένωσης από τις αρχές του 2014. Η Επιτροπή λειτουργήσε σωστά. Στο πλαίσιο του ελέγχου επιλέξαμε και μελετήσαμε τρεις ε, διεθνείς καταστροφές ενώ ε, όπου χρησιμοποιήθηκε ο μηχανισμός. Βοσνία Ζεβοβίνη τον Μάιο του 2014 η επιδημία της έμπολα στη Δυτική Αφρική το Μάρτιο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο 2016 και τον, ο σεισμός στο Νεπάλ τον Απρίλιο του 2015. Σε κάθε μία από αυτές τις καταστροφές η ενεργοποίηση του UCPM έγινε εγκαίρως και η χρήση των ομάδων πολιτικής προστασίας και η διευκόλυνση του συντονισμού στο επιτόπου με συμμετέχουσες ομάδες η διευκόλυνση ενισχύεται με την διάδοση των πληροφοριών, η επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα της Κομισιόν και με, άλλα, ε, με άλλους φορείς ε, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πολλές φορές τα Ηνωμένα Έθνη είναι αυτά τα οποία καθοδηγούν την ομαλή μετάβαση. Φυσικά, όπως είπαμε και την έκθεση, πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και όσον αφορά τη λειτουργία του UCPM, το δικαστήριο από τις λεπτομέρειες της εργασίας του βρήκε, βρήκε κάποια σημεία όπου χρειάζεται περισσότερη προσοχή στις λεπτομέρειες. Με δύο λόγια, οι συστάσεις μας αφορούν το χρόνο, κάποια χαρακτηριστικά του συστήματος ενημέρωσης, στοιχεία του συντονισμού στο πεδίο και την ανάπτυξη και την, υποβολή, και την υποβολή αναφορών. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις μικρές αυτές αλλαγές θα ενισχύσει έτσι περαιτέρω την αποτελεσματικότητα του πολύτιμου αυτού εργαλείου για να μπορέσει την Ένωση, η Ένωση και τα κράτη-μέλη να είναι έτοιμα να ανταποκριθούν σε καταστροφές οπουδήποτε και οποτεδήποτε και αν προκύψουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Κάντεμπαχ. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω θερμός ε, ως εισηγήτρια. Πάντοτε χαίρομαι όταν έρχεται κάποιος από το ελεγκτικό συνέδριο και μας παρουσιάζει μια ειδική έκθεση που ουσιαστικά λέει ότι η δουλειά έγινε πάρα πολύ καλά ε, και ότι ο μηχανισμός στην προκειμένη περίπτωση πολιτικής προστασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λειτουργεί, είναι πλήρως επιχειρησιακός. Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω όλος ιδιαίτερος είναι η τιμότητα και η προθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις ε, και να εφαρμόζει τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Είναι σημαντικό εδώ να υπάρξει μια γρήγορη συντονισμένη δουλειά γιατί αυτές τις επιπτώσεις ε, τις είδαμε και τους τελευταίους μήνες και εβδομάδες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν υπάρχει ταχεία συντονισμένη δράση μπορούμε να γλιτώσουμε τον κόσμο από βάσανα και από πολλή ζημία και βλάκλος να την περιορίσουμε. Συγγνώμη που χτυπάει και το κινητό μου. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την Κομισιόν στις προσπάθειές της, πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι πόροι και οικονομικοί μεταξύ άλλων και βέβαια θα πρέπει να κινητοποιηθούν περισσότερο οι εμπειρογνώμονες, ώστε οι πληγήσεις χώρες ε, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να στηρίζονται και επίσης ε, τονίζουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα σημεία εστίασης ε, επιτόπου για την πολιτική προστασία. Υπήρχε ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που θέλω να ε, αναφέρω. Το 2016, το Φεβράριο, ε, άρχισε να λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα, το οποίο ουσιαστικά ενισχύει αυτές τις θελοντικές δεξαμενές, τις θελοντικές ομάδες και αυτό σχετίζεται με την κρίση έμπολα, δαντλήθηκαν τα διδάγματα. Πάντοτε αυτό το, και ισχύει αυτό παντού. <clears throat> είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει άσκοπη, ε, δεν πρέπει να υπάρχει άσκοπο άχθος ε, διοικητικό γιατί ιδίω ε, εν και το πόσο χρονοβόρες μπορεί να είναι αυτές οι διαδικασίες, ε, το θέμα είναι ότι υπάρχουν καθυστερήσεις που εμποδίζουν και τα κράτη-μέλη αλλά ε, και το κέντρο για τον έλεγχο και την πρόληψη των κρίσεων. Μία παράκληση να υπογραμμίσουμε για τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη κυρίως να προβλέψουν περισσότερους πόρους όχι μόνο οικονομικούς αλλά και ανθρώπινους ε, και τεχνικούς ε, για αυτές τις ελληνικέ ομάδες ώστε να υπάρχει ε, μεγαλύτερη τιμότητα αντίδρασης στις καταστροφές. Ένα θερμό ευχαριστώ και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, που φαίνεται να λειτουργεί κατά το μάλλον ήτον θετικά. Υπάρχει αυτό το σύστημα εσωτερική συνεργασία. και θέλω να πω εδώ ότι και εμείς ε, οι βουλευτές ε, μπορέσαμε να ε, δούμε πόσο καλά λειτουργεί το ERCC. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία αλλά το βασικό είναι ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και επίσης επαναλαμβάνω ότι η Κομισιόν δείχνει την προθυμία να εφαρμόσει πολύ γρήγορα τη συστάση. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλέ υποθέσει που λήγουν. Ε, αυτό το οποίο απαιτείται σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση είναι ώστε να το πιο ταχεία δράση. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, πραγματικά ενδιαφέρουσα ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου με παραδείγματα που μας βοηθούν πολύ και εμεί έχουμε πάει πολλές φορές επί τόπου ε, έχουμε δει τι γίνεται με τις φυσικές καταστροφές και πώς αντιμετωπίζονται ένας τομέας ε, που έχει ήδη πολλή εμπειρία κομισιών. Ο συνάδελφος Αλαφράγκα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μας ε, για την έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου και για το έγγραφο εργασία της εισηγήτριας. Αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργήσε αποτελεσματικά για να διευκολύνει το συντονισμό ε, των αντιδράσεων. Αυτό ήταν ε, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση αυτή, όμως ε, υπάρχει ένα ακόμη πιο σημαντικό τμήμα του προπολογισμού που αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρεις καταστροφές ε, που αναλύθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο, η ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας ε, διευκόλυνε το συντονισμό επιτόπου με τις ομάδες των κρατών μελών. Υιοθετήθηκε ε, μια ολοκληρωμένη εστίαση από την πλευρά της Κομισιόν. Η Κομισιόν κατέβαλε περαιτέρω προσπάθειες μέχρι να ενεργοποιηθούν οι απαντήσεις, οι αντιδράσεις, ε, αν και η ανάπτυξη αυτού του μηχανισμού ήταν αργή. Όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή υπάρχει και εδώ περιθώριο βελτίωσης ε, και αυτό αφορά την ταχύτητα των επεμβάσεων. Ήταν αποτελεσματικέ, αλλά θα μπορούσαν να δοθούν περαιτέρω κίνητρα. Μπορούμε να βελτιώσουμε και τις ε, διαδικασίες ενεργοποίησης κονδυλίων αλλά και εμπειρογνωμόνων επιτόπου, όπως είπε, η συγκήτρια να καταργήσουμε το διοικητικό άχθος, ε, γιατί χάνουμε περαιτέρω χρόνο, να συνεχίσουμε με την ανταλλαγή πληροφοριών με τα Ηνωμένα Έθνη και με τα κράτη-μέλη που είναι κύριοι πρωταγωνιστές ε, ε, σε αυτό το πλαίσιο των φυσικών καταστροφών, αλλά και να ενεργήσουμε έτσι ώστε ο μηχανισμός στο πλαίσιο της πρόληψης να μπορεί να λειτουργεί. Έτσι λοιπόν, ε, Πρόεδρε, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για μια δουλειά που κάνει καλά η Κομισιόν, για το έγγραφο τη εισηγήτρια και την έκθεση του λεκτικού συνεδρίου. Αλλά, αν και όλα αυτά είναι πολύ ικανοποιητικά, να δούμε πώ μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σφαρή, ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν ε, και αυτό το η έκθεση ασχολείται με καταστροφές εκτός τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω και τις καταστροφές που έγιναν στη χώρα μου τον περασμένο. Τίποτα. Και για να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την εξαιρετική δουλειά συντονισμού στη χώρα μου. 45 λεπτά, συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφε. Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει η διαρμηνία. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Μπορεί να μιλήσει πορτογαλικά ο μιλητής, τώρα λειτουργεί. You are English is audible now. Okay. Uh, um, yeah, if it's a... Ξεκινήστε εκ νέου παρακαλώ. Αν είναι πρόβλημα με τη γλώσσα μπορώ να μιλήσω αγγλικά. Λοιπόν, όπως έλεγα, αν ε, και αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση έχει να κάνει με καταστροφές που έγιναν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που σχετίζεται με αυτές τις καταστροφές. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσα εδώ παρά να τοποθετηθώ και εγώ για την εξαιρετική δουλειά που έκανε η Κομισιόν σε αυτό το τομέα. Και θέλω να πω ότι λίγα λεπτά, 45 λεπτά αφού το κράτος ε, μέλος μου ε, αντέδρωσε η Κομισιόν ε, έστειλε βοήθεια για την κατάσβεση των πυρκαγιών, αυτή την καταστροφή που βιώσαμε τον περασμένο μήνα. Εδώ λοιπόν όταν ε, ασκούμε κριτική ε, στην Κομισιόν το κάνουμε, αλλά όταν πρέπει να επενέσουμε την Κομισιόν για τη δουλειά της πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Ήταν εξαιρετική ε, η δουλειά της Κομισιόν και θέλω να την ευχαριστήσω εξ του λαού μου και πραγματικά μπορέσαμε να σώσουμε πάρα πολλές ζωές με, αυτό το, με αυτή την άσκηση. Παρ' όλα αυτά πέθαναν παρ' όλα αυτά αρκετοί άνθρωποι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ε, αναφορά σε αυτή την ε, εντός ένωσης φυσική καταστροφή. Θέλω να δώσω στον εκπρόσωπο του ΕΚΟ. Φρανς Ντέβις, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι και εγώ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ όταν υπάρχει τόσο θετική ανταπόκριση. Ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, την, την εισηγήτρια και τα επιπλέον σχόλιά τη. Πάντοτε υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Αυτό το παραδεχόμαστε, το έχουμε παραδεχτεί και στην επίσημη απάντησή μα και είμαστε, ε, έχουμε αφοσιωθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε σαφώς διατυπώσει και σκεφτεί ότι ε, αυτό το οποίο κάνουμε, γνωρίζουμε ότι αυτό το οποίο κάνουμε έχει σημασία για ανθρώπους και στην Ευρώπη και εκτός. Ως γραφειοκράτες θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα θα λειτουργεί όσο δεν το πιο αποτελεσματικά και όσο δεν το ταχύτερα. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις στην έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου, από τον οποίο έχουμε ήδη κινηθεί. Ε, θα ήθελα δύο λόγια να πω επ' αυτού. Το πιο σημαντικό όσον αφορά το να κερδιθεί χρόνος στι πρώιμε φάσει της ανταπόκρισης με ή χωρί την εντός ή εκτός Ευρώπης. Σήμερα το πρωί ο Γιάννη Λούχνερ είχε συμμετάσχει σε μια συνεδρία των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Εντέβε που παρουσίαζε τη δουλειά που κάνουμε για να αξιολογούμε τον πλήρη μηχανισμό σε αυτό το ενδιάμεσο σημείο. Η συγκεκριμένη πρόταση του ελεκτικού συνεδρίου μας ε, κινητοποίησε σχετικά με το ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να καταγράφουμε πόσο γρήγορα μπορούμε να δράσουμε. Και είδαμε κάποιες από τις ε, ε, κινητοποίησεις μας, πώς το αναλάβαμε, το ξεκινήσαμε αυτό στο επιχειρησιακό επίπεδο και στον, ε, στον και στο πεδίο. Στην, στη, Στη Χιλή κινητοποιηθήκαμε εντό 48 ώρων, είχαμε ε, ομάδες από την, Ιταλία, από την Ισπανία και τη Γαλλία ε, και μπορέσαμε να είμαστε στο πεδίο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι μόνο ο συντονισμός ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πόσο γρήγορα μπορούν να ανταποκριθούν αυτοί τους οποίους συντονίζουμε. Και επίσης θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για τις ζωές που χάθηκαν στην Πορτογαλία και όσον ευχαριστώ για την αναφορά στην πρόσφατη παρέμβασή μας στην Πορτογαλία. Σήμερα το πρωί μας ζητήθηκε βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης στις 5 και 44 το πρωί στις 18 Ιουνίου μια Κυριακή και όσοι από εσά έχετε ε, επισκεφθεί το κέντρο ε, ε, εκτάκτου ανάγκης που λειτουργεί σε 24 τετράωρη βάση δείχνει ακριβώς την αξία αυτή τη παρακολούθηση, γιατί μέχρι τις 7 το πρωί η γαλλική κυβέρνηση είχε ήδη κάνει την πρώτη προσφορά για πυροσβέστες και μέχρι τις 5.30 ε, η Πορτογαλία είχε ζητήσει επιπλέον βοήθεια και ξέραμε ότι πρέπει να κινηθούμε εξαιρετικά γρήγορα. Μέσα σε μισή ώρα οι Ιταλοί συνάδελφοι είχαν προσφέρει δύο επιπλέον Καναντέρ πυροσβεστικά αεροπλάνα και εντός μιας ώρας οι Ισπανοί συνάδελφοι είχαν και αυτοί προσφέρει επιπλέον δυναμικότητα. Οπότε, εντός της ημέρας, η δυνατότητα πυρόσβεστης από τους γειτονικές χώρες και μέσω της, ε, του μηχανισμού συντονισμού της Ευρώπης έκανε υπερπτήσεις και αντιμετώπιζε τη φωτιά. Πρόκειται για μια σημαντική δραστηριοποίηση. Εμείς από πλευράς μας κάναμε κάτι που έχει επισημανθεί και στην έκθεση και στην έκθεση ε, της εισηγήτριας. Συγκαλέσαμε όλες τις υπηρεσίες και όλους όσοι έπρεπε να παρίστανται την πρώτη ημέρα, ήδη εκείνη την ημέρα σκεφτήκαμε πού θα, πού θα χρειαστεί περισσότερη, ε, χρησιμοποιηθούν περισσότερα μέσα. Θέλω λοιπόν να το υπογραμμίσω αυτό. Επίσης, έχουμε επενδύσει και ε, στις συστάσεις που αφορούν το απότερο μέλλον. Έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη ανάπτυξη του το ΣΕΣΙΣ, του Κοινού Συστήματος Επικοινωνίας και Πληροφοριών, που βοηθά την υποστήριξη των κρατών μελών και την χρήση του συστήματος από αυτά. Άμεσα κινητοποίησαμε μια ομάδα εργασίας των χρηστών, συντάξαμε ένα σχέδιο για να εξασφαλίσουμε ότι τα αιτήματα για χρηματοδότηση μεταφοράς θα μπαίνουν αυτόματα στο σύστημα και αυτό δείχνει πόσο φωσιωμένοι είμαστε στο να εξορθολογήσουμε τις διοικητικές διαδικασίες. Οι γραφειοκράτες δεν θέλουν να δρουν γραφειοκρατικά. Ε, εδώ μελετάμε όσο το δυνατόν γίνεται ε, τρόπους, να βρούμε τρόπους που μπορούμε να εξομαλύνουμε την όλη διαδικασία. Η χρηματοδότηση της μεταφοράς είναι το μεγαλύτερο πεδίο αυτή τη στιγμή, αλλά επίσης εισάγουμε μια, ένα τυποποιημένο σύστημα υποβολής σε όλη την Επιτροπή και για άλλους τομείς που αφορά τα έργα πρόληψης και προετοιμασίας αυτό το κάνουμε φέτο. Επίσης βλέπουμε πώς θα αμείβουμε τους εμπειρογνώμονε που χρησιμοποιούνται στις ομάδες. Είναι πολλά τα διοικητικά κομμάτια, οι διοικητικέ λεπτομέρειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν και άλλα θέματα που επισημάνθηκαν από την έκθεση. Δεν θα υπησέλθω στις λεπτομέρειες, δεν ξέρω ότι ήδη έχετε κουραστεί, ε, αλλά πράγματι πρέπει να σα πω ότι έχουμε πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον για τη δουλειά μας και έχουμε κατά νου να σχεδιάσουμε αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε τώρα και αυτά τα οποία ενδεχομένως θα πρέπει να να μας οδηγήσουν σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος της νομοθετικής περίοδου για πιο θεμελιώδεις αλλαγές. Θα επανέλθουμε στο Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο ή, εν πάση περιπτώσει, το φθινόπωρο για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Βέσπερκ, για να κλείσουμε. Έχετε να σχολιάσετε κάτι? Κοιτάξτε, δεν έχω ιδιαίτερα σχόλια, ίσως ένα. Εδώ και έξι χρόνια εργάζομαι στις εξωτερικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι μία από αυτές. Έχω δει πολλά προβλήματα με το συντονισμό. Ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχω δει σε όλες μου τις εκθέσεις. Αυτό είναι το κύριο παράδειγμα του αντιθέτου. Όπως ο συντονισμός ε, λειτουργεί πολύ ομαλά έτσι λοιπόν θα ήταν καλό να δούμε γιατί στην περίπτωση αυτή λειτουργεί τόσο καλά ο συντονισμό ενώ δεν λειτουργεί τόσο καλά σε άλλου ε, τομεί ε, που αφορούν τι εξωτερικέ δραστηριότητε. Ευχαριστώ. <laughs> Είδαμε ένα παράδειγμα καλής πρακτικής σήμερα. Λοιπόν, ε, κυρία Κάντμακ, ε, με δύο προτάσεις. Πάντα αυτά θέλω από το ελεκτικό συνέδριο, είτε κανονικέ είτε ειδικέ εκθέσεις που δεν θα πρέπει να μας απασχολούν ε, σε σχέση με το τι μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά να μπορούμε να τις καταχωρήσουμε ως ευέλτιστες πρακτικές. Γιατί αυτό συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των θεσμικών οργάνων, αλλά και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευχαριστώ πολύ. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρωινή συνεδρίαση. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς που έδωσαν ένα παραπάνω περιθώριο. Έχουμε στις, 12, στις 2.30 ένα ε, θέμα χωρίς διερμηνία. Ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δράση, Δράσης, πώς διαχειρίζει τα κτίρια της ανά τον κόσμο και θέλουμε να δούμε τι γίνεται με τα γραφεία στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον που είναι υπερβολικά ε, ευρύ χώρα, θα έλεγα με πολύ μεγάλη χώρα. Αυτά θα τα πούμε χωρίς δερμία στις